Hölgyeim és Uraim, jó reggelt kívánok! Kálimera, κυρίες ki, kéri. Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm mindannyiukat, és megnyitom. Καλημέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να κηρύξω την έναρξη της σημερινής μας συνεδρίασης. Έχουμε ε, κάποια σημεία στην ημερήσια διάταξη που αφορούν ε, διερευνητικές ε, αποστολές που πραγματοποίησαμε πέρυσι. Η πρώτη ήταν η επίσκεψη στο Λονδίνο ε, για τις υιοθεσίε, αν θυμάστε. Η σχετική αναφορά υπευλήθη, συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη μετά από αίτημα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Βλέπω ότι η κυρία Μίτση μόλις ήρθε. Λοιπόν, η συνάδελφος η κυρία Μίτσι θέλει κανένα δύο λεπτά να καθίσει και στο μεταξύ θα δώσω το λόγο στην κυρία Ταραγώνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μας αναλύσει τη σχετική αναφορά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ονομάζομαι Μάρτα Ταραγώνα Φενόσα και Εργάζομαι στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης Τμάνι Λίκων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον που δείξατε να δώσετε μια συνέχεια στην διαρευνητική αποστολή που πραγματοποιήσατε στο Ηνωμένο Βασίλειο για το θέμα τη υιοθεσία χωρί συνένεση. Όπω είπε ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα σε ουσιαστικό οικογενειακό δίκαιο, ούτε για το ρόλο των ε, φορέων και αρχών προστασία ανηλίκων ή κοινωνική προστασία. Η θεσία διέπεται από εθνικές διατάξεις και κάποιες διεθνείς συμβάσεις. Δυνάμει των συνθηκών, των ευρωπαϊκών συνθηκών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει γενικέ αρμοδιότητες για να παρέμβει στα κράτη-μέλη. Μπορεί να το κάνει μόνο σε περίπτωση που εμπλέκεται τμήμα ενωσιακού ή διάταξη ενωσιακού δικαίου. Για την εθεσία λαμβάνεται υπόψη το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού. Αυτό είναι το πρωτορχικό κριτήριο δυνάμει του άρθρο 21 τη σύμβαση στο ΙΕ για τα δικαιώματα των παιδιών στο, στην οποία συμβαλωμένα μέρη είναι όλα τα κράτη-μέλη. Βέβαια, τα διεθνή πρότυπα δεν αποκλεί το θέμα της υιοθεσίας. Η υιοθεσία χωρίς ε, συνένεση του γονέα υπάρχει, προβλέπεται. Μπορεί να μην είναι το καλύτερη, η καλύτερη λύση για τα παιδιά, αλλά η ανάλυση του υπέρτερου συμφέροντος θα πρέπει να γίνει περιπτωσιολογικά και φυσικά θα πρέπει να γίνει ακρόαση και με τον ανήλικο σε περίπτωση υιοθεσία χωρί την συνένεση του βιολογικού γονέα, να πάκεται στα κράτη-μέλη και τι δικαστικέ αρχέ να εξακριβώσουν ε, το σεβασμό και την τήρηση των δικαιωμάτων των παιδιών με βάση την εθνική νομοθεσία και τις ε, διεθνείς υποχρεώσεις ε, από τις διεθνείς συνθήκες. Σε ό,τι φορά ένα διασυνοριακό στοιχείο, ο κανονισμός 2221 του 2003 ο κανονισμό Βρυξέλλες 2 που βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρηση, αφορά μόνο το ζήτημα δικαιοδοσία για την αναγνώριση και επιβολή δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν σε άλλη χώρα μέλος. Και αυτό αφορά το άρθρο 56 ε, που αποκλεί όμω την υιοθεσία από το ουσιαστικό πεδίο εφαρμογή του κανονισμού. Απλώ αφορά την ε, θέση ενό παιδιού σε άλλο κρατός μέλος. Οπότε το αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απλούστευση των διαδικασιών σε ό,τι αφορά την, ε, ανάθεση ενός παιδιού σε κυδαιμονία σε άλλο κράτος μέλος ε, ελήφθη υπόψη. Παρ' όλα αυτά, η αρμοδιότητα για τη λήψη προστατευτικών μέτρων ε, επαφείται στα κράτη-μέλη, στο οποίο διαμένουν τα παιδιά και ισχύει η εθνική νομοθεσία. Επίσης, όλα τα κρατη το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν προσυπογράψει την ε, σύμβαση του 96 για τα δικαιώματα του παιδιού. Το 7ο, 8ο και 1 το φόρουμ για τα δικαιώματα του παιδιού επικεντρώθηκε σε θέματα συντονισμού και συνεργασίας ε, στα θέματα προστασίας παιδιού με βάση τα διεθνή πρότυπα. Και μάλιστα ε, τα έγγραφα του 1 του φόρουμ περιέλαβαν νέα αρχές για τη συμπερίληψη στα συστήματα προστασίας του παιδιού. Για παράδειγμα, θα πρέπει να ενισχυθούν τα προληπτικά μέτρα προκειμένου να απαφευθεί στο μέτρο του δυνατού. Συμπεριλαμβανομένου του χωρισμού του παιδιού από τους γονείς. Και επίσης ε, ζητούμε συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των συστημάτων προστασίας των παιδιών. Προσφάτως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια αφαίρεσε κάποια κονδύλια για την ενίσχυση της δικαστικής εξουσίας και την κατάρτιση ε, για τέτοια θέματα. Σε ό,τι αφορά τις ε, χρηματοδοτικές μας προτεραιότητες, λαμβάνουμε υπόψη τα διεθνή πρότυπα προκειμένου να γίνει μια καλύτερη ολοκλήρωση και συντονισμό των διαφόρων εθνικών συστημάτων προστασία των παιδιών. Ευχαριστούμε. Και θα ήθελα να ακούσω του συναδέλφου που θέλουν το λόγο. Κυρία Μίτση, πρώτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Καυτό το θέμα που προκαλεί και πολλά έντονα συναισθήματα ε, για όσους επισκέφθηκαν το Λονδίνο κιόλα, εγώ πριν από μερικά χρόνια και φάνηκε ότι είναι πολλά τα προβλήματα που πρέπει να λυθούν και ξεπερνούν το συναισθηματισμό αγγίζουν πολλά, πολλά θέματα πολλά, πολλούς τομείς Γι' αυτό ήθελα να δω τι θα μας πει η Επιτροπή. Ε, με απασχολεί αν έχετε καθόλου δεδομένα, στατιστικά δεδομένα, μια καλύτερη συνολική εικόνα για το τι γίνεται όχι μόνο για τις μη συνενετικές υιοθετησίες σε εθνικό επίπεδο, αλλά και γενικότερα το δίκαιο το οικογενειακό που επιτρέπει να γίνουν σωστές συγκρίσεις μεταξύ των νομοθεσιών των κρατών μελών. Επίσης με απασχολεί κατά πόσον η Επιτροπή έχει πληροφορίες ότι τα εθνικά δικαστήρια για το οικογενειακό δίκαιο συστηματικά εφαρμόζουν τη σύμβαση της Βιέννης στην αρχική φάση της ε, ανάθεσης δημονίας των παιδιών και εάν εκπροσωπούνται σωστά οι διάδικοι για τις διασυνοριακές υποθέσεις εφόσον πρόκειται για περιπτώσεις μεικτών υποθέσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει καθόλου πρωτοβουλίε όπω σύστησε η Επιτροπή μα για να εκπονήσει συγκεκριμένε κατευθυντήριε γραμμέ για το συντονισμό και τη συνεργασία και την, ε, τα σφαιρικά συστήματα προστασία των παιδιών που θα λαμβάνουν σε κάθε φάση τη διαδικασία υπόψη τι ανάγκε του παιδιού για προστασία και θα παρέχουν τι σχετικέ υπηρεσίε. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι. Άλλος, κανείς. Παρακαλώ κυρία Ταραγώνα Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και κυρία Μίτση για τις ερωτήσεις σας. Δυστυχώς όπως ε, ε, αφού οι συναδελφοί που ασχολούνται με τα θέματα αυτά κολλείονται σήμερα θα διαβιβάσω τα ερωτήματά σας και θα σας απαντήσουν γραπτός. Όσον αφορά το τελευταίο ερώτημα για ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας ε, παιδιών. Σας ε, παραπέμπω στα όσα είπα προηγουμένως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, thank ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Μίτση. Τι προτείνετε να κάνουμε, να το κρατήσουμε ανοιχτό και να περιμένουμε. Ναι, ναι κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά για να μας δώσει μια ικανοποιητική απάντηση η Κομισιόν. Συμφωνείτε όλοι? Ωραία. Ωραία, το κρατάμε ανοιχτό και περιμένουμε. Το δεύτερο θέμα στην ημερήσια διάταξη σχετίζεται με την επίσκεψή μας στην Ισπανία και το σχετικό έγγραφο βεβαίως την έκθεση για τους ποταμούς Εύρω και Ταχώ και την χρήση των υδάτων τους. Ε, εγώ ήμουν μάλιστα επικεφαλής ε, της αντιπροσωπείας για την επίσκεψη αυτή το 2016. Είχαμε έναν δομημένο διάλογο μετά εδώ στην Επιτροπή μας. Θεωρώ ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή έκθεση η Ισπανική κυβέρνηση έκανε κάποια βήματα μετά από αυτήν την έκθεση και μάλιστα προχτές ήδη διαπιστώσαμε ότι η Κομισιόν είχε κινήσει διαδικασίες κατά της Ισπανίας γιατί η Ισπανία δεν είχε αναλάβει όλες τις απαιτούμενες δράσεις. Οπότε μιλάμε για ένα σημαντικό διάλογο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ισπανικού κράτους. Λοιπόν, η πράσινη είχαν ζητήσει να μπει το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη και θα τους δώσω τον λόγο. Αλλά πρώτα θα στραφώ στην κυρία Ελίζα Βάργκας Αμεγίν που εκπροσωπεί την Κομισιόν. Μπορείτε να μας πείτε λοιπόν τι συμβαίνει. Συγγνώμη, λάθος. Ε, είναι εδώ και οι αναφέροντες από την Ισπανία Χώνα Μογκρέσπο Αγκουγιάρ και Μαντήλ Φροντέν έχετε τον λόγο για 5 λεπτά και με συγχωρείτε Σας ευχαριστώ Καταρχήν δεν το γνωρίζαμε αυτό κύριε Σάκη ε, άρχισε η εκπόνηση έκθεση. Δεν είχαμε ιδέα για αυτό που είπε ο πρόεδρο. Θα σα εκφράσουμε απλώ τη δική μα άποψη για το θέμα. Κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, η πλατφόρμα για την προάσπιση του εύρου είναι ένα οριζόντιο κοινωνικό κίνημα. Η μοναδική μα αξίωση είναι να προστατεύσουμε τον ποταμό Εύρο και το δέλτα του Εύρου, γιατί είναι ο τρίτο σημαντικότερο υγρότοπο τη Μεσογείου, μετά το δέλτα του Νείλου και την Γαλλική Καμάργ. Το δέλτα του Εύρου είναι 320 τετραγωνικά χιλιόμετρα με υψηλή οικολογική αξία. Είναι στρατηγικό τόπο για τι μεταναστευτικέ κινήσει των αποδημητικών πτηνών μεταξύ Αφρική και Ευρώπη. Επιπλέον, 325 είδη πτηνών βρίσκονται στο Δέλτα από τα 600 είδη που υπάρχουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι λοιπόν τόσο σημαντικό για τη βιοπικιλότητα του Δέλτα του Εύρου, και γι' αυτό εμπίπτει σε όλες τις μορφές διεθνού προστασίας που υπάρχουν. Είναι ζώνη Ράμσαρ, ζώνη ΣΕΠΑ, ΛΙΚ, με βάση το δίκτυο Natura 2000 και από το 2013 είναι και ειδικού προστατευμένη ζώνη της βιόσφαιρας της UNESCO. Επίση υπάρχει μεγάλη οικονομική δραστηριότητα γύρω από την γεωργία, κυρίω λόγω τη οριζοκαλλιέργεια. Για να μην μιλήσουμε για την ε, αλία και την ήχθειοκαλλιέργεια, που επίση είναι σημαντικέ. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε και βιώσιμο τουρισμό, περιβαλλοντικό. Γι' αυτό θεωρούμε ότι το, Δέλτα, το Δέλτα του Εύρου είναι ένας ε, ιδιαίτερος τόπος μίζωνος οικολογικής σημασίας, ενώ ταυτόχρονα είναι πολύ εύθραυστο οικοσύστημα και οποιαδήποτε προσβολή μπορεί να το πλήξει ή να το εξαφανίσει. Και μάλιστα όταν έγιναν τα μεγάλα φράγματα στη λεκάνη του ποταμού, η υποχώρηση των ειζημάτων προς το Δέλτα μειώθηκαν κατά 90% γιατί παρέμεναν στα φράγματα αυτά τα ειζήματα. Επίσης είχαμε πολύ σημαντική μείωση των κοιτών των ποταμών, των παραποτάμων του Εύρου. Άρα αυξήθηκε ε, η μόλυνση λόγω της έλλειψης της ε, διάλυσης, της αλλίωσης. Εξαιτής λοιπόν της έλλειψης της μείωσης των και των μικρότερων ε, κοιτών, το Δέλτα εξαφανίζεται χρόνο με το χρόνο. Σήμερα είναι η τέταρτη φορά που ερχόμαστε στην Επιτροπή Αναφορών για να σας παρουσιάσουμε την αναφορά μας. Και συνεχίζουμε να έχουμε το ίδιο αίτημα, γιατί πιστεύουμε ότι κάθε φορά που η Ισπανική κυβέρνηση κάνει ένα νέο υδρολογικό σχέδιο, δεν λαμβάνει υπόψη ούτε προτείνει συγκεκριμένα μέτρα με αποδεδειγμένα επιστημονικά πορίσματα για να προστατεύσει αυτή την ε, ευρωπαϊκή ζώνη μείζωνος περιβαλλοντικής σημασίας, στην οποία διαβιούν χιλιάδες άνθρωποι. Επίσης θεωρούμε ότι η Ισπανική κυβέρνηση δεν έλαβε υπόψη τις συστάσεις της έκθεσης της Επιτροπής ε, ε, Αναφορών του 2016. Το υδρολογικό σχέδιο του Ιανουαρίου του 2016 της Ισπανικής κυβέρνησης εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, που είναι το ελάχιστο σε ό,τι αφορά την οδηγία πλαίσιο για το είδωρ, την οδηγία για τα πτηνά και την οδηγία για τα ενδιατήματα. Το τελευταίο υδρολογικό σχέδιο λοιπόν εξακολουθεί να είναι πιστή αντιγραφή του προηγούμενου χαλκομανία του προηγούμενου. Και θεωρούμε ότι το νέο υδρολογικό σχέδιο θα επιδεινώσει τα προβλήματα που σας περιέγραψα. Γιατί συνεχίζει να προτείνει 420.000 νέων αρδεύσιμων καλλιεργειών και επίσης 59 καινούργια φράγματα σε όλη τη λεκάνη απορροής του Εύρου. Στη λεκάνη απορροής του Εύρου Ήδη έχουμε τα περισσότερα φράγματα από όλα τα ευρωπαϊκά ποτάμια, γύρω στα 200 φράγματα. Γι' αυτό λοιπόν, αν το νέο υδρολογικό σχέδιο υλοποιηθεί, θα οξύνει ακόμη περισσότερο το πρόβλημα της συγκράτησης των ειζημάτων στα φράγματα. Έτσι, θα έχουμε μείωση του φυτοπλακτών προς την θάλασσα και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την αλία και για την ηχθειοκαλλιέργεια που είναι σημαντικό, σημαντική πηγή πλούτου και οικονομική και περιβαλλοντική. Ήδη σχετικέ οικονομικέ δραστηριότητε επλήγησαν τι τελευταίε δεκαετίε, αλλά μπορούν να επιδεινωθούν ακόμη περισσότερο τα προβλήματα. Μελέτε δείχνουν την αιτιώδη σχέση μεταξύ των αλλιευμάτων και των μαλακίων από τον Εύρο που φτάνουν ε, στη θάλασσα. Επίση, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ε, διείσδυση ε, αλάτινο ύδατο στα υπόγεια ύδατα. Έτσι, ίσω τροποποιηθούν τα ντόπια είδη που δεν αντέχουν το αλατισμένο νερό. Και γι' αυτό ήδη έχουμε 30 χιλιόμετρα νερού θαλάσσιου μέσα στη, στο γλυκό νερό του ποταμού. Και μάλιστα αναμένω ότι θα φτάσει στα 50 χιλιόμετρα διείσδυση του, του θαλάσσινου νερού στο ποτάμιο. Θέλουμε λοιπόν ένα νέο καθεστώς που θα εξασφαλίζει την προστασία αυτού του στρατηγικής σημασίας ε, υγροτόπου για την χλωρίδα και την πανίδα. Πολλές μελέτες έχουν γίνει για το Δέλτα του Εύρω, αλλά χρειάζονται και άλλες για να δούμε τι μέτρα χρειάζονται για να παρεμποδιστεί η περαιτέρω ε, διάβρωση του Δέλτα και μάλιστα να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση. Θα πρέπει να περιοριστεί ο αριθμό των φραγμάτων και των αρδεύσιμων καλλιεργιών. Αλλά δεν είναι αυτό ο καλύτερο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του ΔΕΛΤΑ, που είναι γνωστά εδώ και πολλά χρόνια. Όπω αναφέρεται στο σημείο 2 των συστάσεων τη έκθεση τη επιτροπή Αναφορών του 2016, αναφέρονται όλα αυτά. Άλλε συστάσει που είχε η έκθεση επιτροπή Αναφορών ήταν η εξή. Στο σημείο 5 αναφερόταν ότι οι Ισπανικέ αρχέ θα πρέπει να συνεργαστούν με την κοινωνία των πολιτών και μη κυβερνητικέ οργανώσει κατά την εκπόνηση και κατάρτιση των υδρολογικών σχεδίων. Ελάχιστα όμως έχουν αλλάξει από αυτήν την άποψη στη στάση της ισπανικής κυβέρνησης. Η κυβέρνηση συνεχίζει τα γνωστά, τα, τη μέχρι τώρα στάση της, αγνοώντας σε μεγάλο βαθμό την ε, δημόσια διαβούλευση που προτείνουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες και τη γνώμη των ε, ε θυγωμένων. Επίσης, το σημείο 4 της σύστασης τη επιτροπή της ζητείται επιτήρηση για τον υδρολογικό σχεδιασμό και επίση χρηματοδότηση ανεξάρτητων μελετών για τις ανάγκες του ποταμού Εύρου και του Δέλτα του Εύρου με την πραγματική συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων. Θα θέλαμε να επιμείνουμε σε αυτές τις δύο συστάσεις, γιατί επιτέλους είναι και η ώρα για να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα θέματα του εύρου. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια που επιδεινώνεται η κατάσταση, ενώ οι ισπανικές κυβερνήσεις προτείνουν σχέδια διαχείρισης απορροής λεκάνης που δεν προσφέρουν τίποτα καινούριο. Και όπως αναφέρεται στο σημείο 10 των συστάσεών σας, ήρθε η ώρα να εξυγχρονιστεί ο τρόπος προγραμματισμού των υδρολογικών σχεδίων της Ισπανίας. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, σας ευχαριστούμε και πάλι που μας επιτρέψατε να έρθουμε εδώ η πλατφόρμα της προάσπισης του Δέλτα του Εύρου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ελπίζουμε να συνεχίσετε να μας λαμβάνετε υπόψη και στο μέλλον. Μην αρχιοθετήσετε την ε, αναφορά μας θα πρέπει να κάνετε ό,τι μπορείτε ώστε η Ισπανική κυβέρνηση να τηρήσει τι υποχρεώσει τη που απορρέουν από τι ευρωπαϊκέ οδηγίε. Γιατί σε τελική ανάλυση συμμετείχε και η κυβέρνηση στην έγκριση των οδηγιών. Δεν νομίζουμε ότι είναι τίποτα φοβερό αυτό που ζητάει η αναφορά μα. Απλώ ζητούμε να τηρηθούν οι διατάξει και κατευθυντήρε γραμμέ που απορρέουν από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Επίση, οι πολίτες των παρόχθιων περιοχών του εύρου είναι έτοιμοι να μιλήσουν με τον οποιοδήποτε για οποιοδήποτε υδρολογικό σχέδιο, ώστε να βελτιωθεί το Δέλτα του Εύρου ω ζώνη ε, στρατηγική βιοπικιλότητα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ναι, η συνάδελφό σα. Ο κύριος Αγγιλάρ. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. 8 ε, με 10 Φεβρουαρίου του 2016 η Επιτροπή Αναφορών ζήτησε διερευνητική αποστολή στην Ισπανία για να διερευνήσει την αθέτηση των υποχρεώσεων της Ισπανικής κυβέρνησης που απορρέουν από την οδηγία πλαίσιο για το είδωρ σε ό,τι αφορά τις λεκάνες απορροής του Εύρου και του Τάγου. Ε, εκ μέρους του ΓΚΟΕ, ε, της ΓΚΟΕ θα ήθελα να σας μιλήσω για την αναφορά 834 του 2012 έγιναν 13 συστάσεις μετά από την διερευνητική αποστολή. Πολλές αφορούν τον τάγο. Θα πρέπει ε, να εξακριβωθεί κατά πόσο τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις και οι δεσμεύσεις της ισπανικής κυβέρνησης. Μάλιστα το υδρολογικό σχέδιο που ήταν το νέο για το 2015-2021, τη 1 η Ιανουαρίου του 2006, είναι πιστή αντιγραφή του προηγούμενου υδρολογικού σχεδίου. Δεν ελήφθησαν υπόψη οι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βελτίωση του πρώτου σχεδίου διαχείρισης τη λεκάνης απορροής για, για καλύτερο υπολογισμό, εξακρίβωση της στήριξης περιβαλλοντικών ε, κριτηρίων, στόχοι των προστατευόμενων περιοχών και ούτω καθεξής. Εμείς θα επικεντρωθούμε σε δύο παραβιάσεις που είναι οι πιο σοβαρές. Την οικολογική ροή και την ανάκτηση του κόστους. Σε ό,τι αφορά την οικολογική ροή του ποταμού, όπως είπαμε, το δεύτερο σχέδιο είναι χαλκομανία του πρώτου σχεδίου υδρολογικού. Δεν έγινε καμία προσαρμογή ε, με βάση τις συστάσεις που έγιναν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Επίσης, ε, η οικολογική ροή θα πρέπει να είναι επαρκής ώστε να συντηρηθούν οι κότοποι και οι προστατευόμενες περιοχές του Natura 2000. Η οικολογική ροή ποταμού δεν αφορά μόνο την ποσότητα του νερού, αλλά και την ε, κατάλληλη χημική σύσταση και την ε, ανάγκη να υπάρχουν διαφοροποίησεις, διακοιμάνσεις ε, στη ροή του ποταμού. Επίσης, ε, θα χρειάζονται μελέτες για να αναγνωριστούν οι πραγματικές ανάγκες ε, των περιοχών σε ό,τι αφορά την ποιότητα του ύδατος και τις οικολογικές ουρές. Μάλιστα και οι αναφερόμενοι και οι τοπικές ε, οργανώσεις και η κοινωνία των πολιτών ζήτησαν να αναθεωρηθεί ε, το υδρολογικό σχέδιο με βάση το άρθρο 14 της Οδηγίας Πλαίσιο. Γιατί έχουμε κακή οικολογική κατάσταση αυτή τη στιγμή που μας απομακρύνουν από την υλοποίηση των στόχων της Οδηγίας. Έχουμε είδωρ κακής ποιότητας που διατηρεί την ίδια ροή ποταμού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και ως εκ τούτου έχει αρνητική επιρροή και στα ενδιατήματα και στα διάφορα είδη που εκεί κατοικούν. Επίση, παραβιάζεται η οδηγία για, τα, για την άγρια πανίδα των πτηνών και η οδηγία για τα διάφορα μέρη του Natura 2000. Το ίδιο ισχύει και για την ανάκτηση του κόστου. Στο άρθρο 9, η οδηγία πλαίσιο για το είδωρο λέει ότι τα κράτη-μέλη θα λαμβάνουν υπόψη την αρχή τη ανάκτηση του κόστου των υπηρεσιών που αφορούν το είδωρο, Ακόμη και το περιβαλλοντικό κόστο που αφορά του σπόρου. Επίσης έχουμε την, το φράγμα του Τάγο και του παραποτάμου Σεγούρα. Είναι ο χειρότερος παράγοντας που συνέβαλε στην επιδίνωση της κατάστασης στον Τάγο. Αυτή, αυτό το φράγμα του Τάγο Σεγούρα στηρίχθηκε σε ένα μοντέλο μη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως φάνηκε την τελευταία τεσσαρακονταετία στην Ισπανία. Οι προηγούμενε κυβερνήσει και οι σημερινοί πρόθεσαν ένα οικονομικό μοντέλο στην ανατολική πλευρά της Ισπανίας που χαρακτηριστικό είναι η λειψιδρία που στηρίζεται σε ένα μη βιώσιμο οικονομικό μοντέλο που στηρίζεται περισσότερο στην πολεοδομική ανάπτυξη, στην εντατική άρδευση και στον τουρισμό με υψηλή κατανάλωση ύδατος. Δηλαδή δημιουργήθηκε ένα τέρας που κατασ... κατασπαθίζει εκατοντάδες τόνους κυβικά μέτρα νερού που είναι ένα σπάνιος πλούτος για την ε, περιοχή. Επίσης ε, μειώνεται η του τάγου. Το μοντέλο αυτό μπορεί να στηριχθεί μόνο στην αφαλάτωση ή στα φράγματα. Ε, δυστυχώς ε, και οι δύο λύσεις είναι δαπανηρές, γιατί η, η αφαλάτωση έχει πολύ ψηλότερο κόστος από τα φράγματα. Ε, γιατί τα φράγματα ε, χρηματοδοτούνται. Οπότε οι Ισπανικές αρχές δεν σέβονται την αρχή της ανάκτησης του κόστους. Το κόστος ε, του ύδατος ε, είναι ένα, το 1 τεσσαρακοστό από το αρχικό κόστος και ένα πεντηκοστό μικρότερο από το κόστος που ε, καταβάλλονται από τις αγορές ε, για, στην περίπτωση της ξηρασίας του 2018. Επίσης, θα πρέπει να πληρώνεται η πραγματική τιμή για το νερό, αλλά τα εμποροκρατικά συμφέροντα και τα οικονομικά συμφέροντα λόγω της ε, ε, του φράγματος και της, ε, με, του φράγματος σε Σεγούρα-Τάγο έχουμε ουσιαστικά διασπάθηση των υδάτινων πόρων χωρίς κανένα ε, έλεγχο περιβαλλοντικής επίπτωσης. Ήδη είχαμε μείωση κατά 48% των υδάτινων πόρων που υπάρχουν ανάντι του τάγου. Και μάλιστα έγινε το φράγμα με σφαλμένους υπολογισμούς και με βάση με τις προβλέψεις αυτές, οι υδάτινοι πόροι ανάντι του τάγου θα μειωθούν ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Η κατάσταση αυτή έχει όχι μόνο αρνητικέ περιβαλλοντικές συνέπειες, αλλά και ε, κοινωνικο-οικονομικές, πολιτισμικές και συνέπειες στο τοπίο ανάντι του τάγου. Στο Αραχουέτ, στο, Τουλέδο, στο Τολέδο και στην Ταλαβέρα ε, και μάλιστα ε, πόλεις που είναι πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO και ο τάγος είναι πολιτιστική κληρονομιά, το τοπίο ε, καταστρέφεται. Έχουμε επίση και τι κλιματικέ αλλαγέ. Ούτε αυτέ ελήφθησαν υπόψη. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την κατάσταση αυτή ω έχει. Ούτε να παραμείνουμε στο δεύτερο αναθεωρημένο σχέδιο για, τον, για την περίοδο 2015-2021 οι Ισπανικέ αρχέ δεν κατάφεραν να τηρήσουν τι συστάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό θα παρακαλούσα να μην αρχιοθετήσετε την αναφορά μα να την κρατήσετε ανοιχτή, πολλό δε μάλλον που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκκίνησε διαδικασία επί παραβάση κατά τη ισπανική κυβέρνηση. Θα πρέπει λοιπόν να παραμείνει εκρεμή η αναφορά, προκειμένου να εξεταστεί ο βαθμό συμμόρφωση τη ισπανική κυβέρνηση με τι κοινοτικέ οδηγίε. Επίση θα πρέπει να γίνει ε, καθαρισμός των λιμάτων, ιδιαίτερα από το παραποτάμους του τάγου. Αν δεν, του τάγου. Αν δεν γίνει τέτοια, τέτοιος καθαρισμός, δεν πρόκειται να βελτιωθεί η περιβαλλοντική κατάσταση του τάγου. Ευχαριστώ. Να σας ενημερώσω ότι υπάρχει και μια μελέτη για την διαχείριση των υδάτων των δύο ποταμών και τη λεκάνη απορροή του. Λοιπόν, να δώσω τώρα τον λόγο στην Κομισιόν. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλημέρα σε όλους σας. Ευχαριστώ και τους αναφερόμενους ε, για τις πληροφορίες που μας έδωσαν. Καταρχήν να σας ε, πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υπόψη τις συστάσεις και τα συμπεράσματα ε, της αποστολής σας ε, στον Τάγο και στον Εύρο. Λάβαμε υπόψη ε, τις συστάσεις σας κατά την εκτίμηση της κατάστασης και την αξιολόγηση των τελευταίων ε, σχεδίων διαχείρισης ε, λεκανών απορροής ποταμών της Ισπανικής Κυβέρνησης. Επίσης, αναφέρθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες και παράβαση των οδηγιών αυτών από την Ισπανική Κυβέρνηση. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να δημοσιεύσει τις εκθέσεις για την αξιολόγηση των δεύτερων ευρωπαϊκών υδρολογικών σχεδίων και θα ακολουθήσουν εκθέσεις. Μία αφορά την Ισπανία και εκεί εξετάζουμε τα συστημικά προβλήματα της Ισπανίας και πραγματοποιούμε και συγκεκριμένα σχόλια που αφορούν ιδιαίτερα τις λεκάνες απορροής του Τάγου και του Εύρου που ενδιαφέρουν κυρίως τους υποβάλλοντες ε, την αναφορά. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ο ρόλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, για την αξιολόγηση των ε, υδρολογικών σχεδίων έχει όρια. Εμείς απλώς αξιολογούμε το περιεχόμενο των υδρολογικών σχεδίων και εξετάζουμε κατά πόσο τηρούνται οι υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι οδηγίες και κυρίως η οδηγία πλαίσιο για το είδωρ. Όπως σας ανέφερα, ε, επίκειται η δημοσίευση αυτών των εκθέσεων με συγκεκριμένες παρατηρήσεις και συστάσεις. Μπορώ όμως ήδη να σας ε, να σας αναφέρω ότι δεν τηρήθηκαν ακόμη οι στάσεις του πρώτου κύκλου, όπως φάνηκε και από τα συμπεράσματα της έκθεσης της Επιτροπής Αναφορών. Εξακολουθούν λοιπόν να ισχύουν οι στάσεις μας με βάση το πρώτο σχέδιο. Μετά την αξιολόγηση που κάναμε και τις, τα συμπεράσματα που θα περιλαμβάνουν οι εκθέσεις μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφασίσει ποια είναι η κατάλληλη συνέχεια που θα πρέπει να δοθεί για τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν ή τα ελλείμματα. Θα χρησιμοποιήσουμε πάντα το μέσο για να απαιτήσουμε την τήρηση των περιβαλλοντικών μας στόχων. Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι εκκρεμούν πολλές υποθέσεις στα εθνικά δικαστήρια που έχουν άμεση σχέση με πολλά σημεία των αναφορών. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά δικαστήρια είναι τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα για να εξασφαλίσουν το σεβασμό του ενωσιακού δικαίου και τη σωστή του εφαρμογή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνηθίζει να μην επεμβαίνει σε τέτοια θέματα εφόσον εκκρεμωδικούν υποθέσεις. Περιμένουμε λοιπόν πρώτα την έκδοση δικαστικών αποφάσεων για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Επίσης, θα ήθελα να σας διευκρινίσω ότι η διαδικασία επί παραβάση που ανέφερε ο πρόεδρο προηγουμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη Ισπανική κυβέρνηση αφορούσε την Δονιάνα, το Εθνικό Πάρκο Δονιάνα. Αυτά, ευχαριστώ. ευχαριστώ. Τώρα η κυρία Βαλέρο, η διακεκριμένη συνάδελφος. Ευχαριστώ. Συμμετείχα και εγώ στην ε, διερευνητική των πραγμάτων αποστολή στον Εύρο και στον Τάγο της Ισπανίας. Για τον Τάγο, για παράδειγμα, νομίζω ότι αυτό που είδαμε ήταν ε, από τα χειρότερα που έχουμε δει για τη λεκάνη απορρόφηση ποταμού. Μα ποιο ποταμό! Δεν υπήρχε καν ποταμός. Στην Ταλαβέρα Δελαρέινα, αυτό που φαινόταν ως ποταμό ε, ποταμός ε, μεγάλος, ουσιαστικά είχαν απομείνει 10-15 εκατοστά ε, νερού στην Κίτη. Υπάρχουν ε, τεράστια προβλήματα. Και στον Τάγο βρισκόμαστε ήδη πρωτοτελεσμένο γεγονότο. Έχει καταστραφεί πια ο Τάγο. Δεν ξέρω πώ θα μπορέσουμε να αντιστρέψουμε αυτή τη διαδικασία και να ανακτήσουμε την κήτη του Τάγου. Και πολύ φοβάμαι ότι και στον Εύρο το ίδιο θα συμβεί. Θα πρέπει να αποτρέψουμε την ε, επιδείνωση και την καταστροφή του Εύρου, όπως συνέβη με τον Τάγο. Μάλιστα, πέρυσι έγινε και μία δεύτερη αποστολή παρακολούθησης ε, για τον Τάγο και μίλησα με το, τις τοπικές κοινότητες, ζητώντας τη γνώμη τους για την κατάσταση. Και θεωρώ ότι οι συστάσεις που κάναμε από την Επιτροπή Αναφορών όταν ε, μετέβουμε στην περιοχή θα πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη. Δεν ξέρω αν τις γνωρίζει αυτές τις στάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα δώσει κάποια συνέχεια ή θα αναλάβει δράση σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης. Από ό,τι ακούσαμε και από τους υποβάλλοντες στην αναφορά, δεν υπήρξε ιδιαίτερη δραστηριοποίηση, καμία διόρθωση. Αναμένουμε τις εκθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μας είπατε ότι όσον όπου θα δημοσιεύθουν. Ναι, αλλά βρισκόμαστε σε στάση αναμονής. Δεν ξέρουμε την άποψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά τις οικολογικές ροές, αυτό είναι πολύ σημαντικό σημείο για τον τάγο, για να επιβιώσει ο τάγος, για να μην εξαφανιστεί τελείως, να μην αποξηρανθεί τελείως. Και το ίδιο ισχύει και για τον Εύρο. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να επέμβετε εφόσον εκκρεμωδικούν υποθέσει στην Ισπανία και περιμένετε την έκδοση των δικαστικών αποφάσεων πρώτα, αλλά αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι πολύ χρονοβόρα. Οπότε, αν καθυστερήσετε ακόμη περισσότερο, η επιδείνωση θα συνεχιστεί. Πιστεύω ότι τώρα θα πρέπει να δράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο είναι καιρό. Γιατί υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος επιδείνωσης της κατάστασης εμείς στις συστάσεις μας ζητήσαμε τη σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής για την αξιολόγηση της κατάστασης. Μια στιγμή να ψάξω τις συστάσεις που κάναμε. Τις ψάχνω αλλά τις βρίσκω. Και να τα πω στα αγγλικά τώρα ζητάει, συνιστά να ξεκινήσει μια ανεξάρτητη εις βάθος μελέτη όσον αφορά την οικολογική επίδραση σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και να δώσει δεδομένα για την αναθεώρηση του επόμενου κύκλου διαχείρισης της λεκάνης απορροής ή δεν ξέρω τι λέει εδώ πέρα και να αποκατασταθούν οι ροές του Δέλτα, του Εύρου και του Τάχο. και πράγματι δεν ξέρω εάν αυτό συνέβη αντιλαμβάνομαι ότι δεν συνέβη οπότε ζητάμε και πάλι συνεργασία συνεργασία με όλους τους διαφορετικούς οργανισμούς και θεσμικά όργανα και βέβαια στην κοινωνία των πολιτών και πέρα από αυτό θυμάμαι πολύ καλά ότι ζητήσαμε από την Ισπανία να αλλάξει κάπως άποψη, να εξυγχρονιστεί στην προσέγγισή της ε, σε ό,τι αφορά τη μεταχείριση των λεκανών απορροής προκειμένου να παραμείνει το νερό στα ποτάμια, να μην οδηγηθούν σε αφανισμό. Τι έγινε. Εξετάσετε αυτά τα θέματα της εκτροπής του Σεγούρα στον Τάγο υπήρξε βούληση της Ισπανικής κυβέρνησης να βελτιωθεί η κατάσταση. Αυτά. Σας ευχαριστώ η Ρόζα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως ο Πρόεδρος Σάκη μίλησε για τη διαδικασία επιπαραβάσει κατά της ε, Ισπανίας για, τις, ε, για τους υδάτινους σπόρους στο Εθνικό Πάρκο της Δονιάνα. Δεν έχουν σχέση με τον Τάγο αυτές οι διαδικασίες επιπαραβάσεις βάρος της Ισπανικής κυβέρνησης. Και εγώ έλαβα μέρος στην αποστολή και είχαμε ε, επαφή και με τους υποβάλλοντες στην αναφορά και με την πλατφόρμα της προστασίας του Τάγου και του Εύρου και με μέλη κυβέρνησης που συμμετείχαν στην εκπόνηση του υδρολογικού σχεδίου για τη διαχείριση των λεκανών απορροής του Τάγου και του Εύρω. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες προβλέπουν τους δύο κύκλους των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής. Ο πρώτος κύκλος ήταν το 2009 με 2015 και ο δεύτερος κύκλος ξεκινά από το 2015 και εκτείνεται μέχρι το 2021. Και μια και το 2009 δεν έγιναν ακόμη τα δεύτερα σχέδια, ουσιαστικά έγιναν ταυτόχρονα τα σχέδια και των δύο κύκλων. Και αυτά τα σχέδια διαχείρισης ε, του Τάγου, του Γουαδιάνα, του Εύρου, του Γουαδαλκιβίρ έτυχαν, την υποστήριξη, έτυχαν της υποστήριξης της Εθνικής Επιτροπής ε, Λεκανών Απορροής. Εκεί συμμετέχουν όλοι οι χρήστες, η αυτόνομη αυτοδιοίκηση και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Το 80% ε, των ε, ενδιαφερομένων ήταν υπέρ της Εθνικής Επιτροπής για τα Υδρολογικά Σχέδια. Επίσης και το Συμβούλιο Επικρατείας της Ισπανίας έδωσε τη θετική του γνώμη και εγκρίθηκε και από το Συμβούλιο Υπουργών. Δηλαδή η συμμετοχή ε, και η διαβούλευση ήταν ε, ευρύτατη. Συμμετείχαν περιβαλλοντικές οργανώσεις, κοινωνία των πολιτών, οικονομικές οργανώσεις και κατά 80% ε, υπήρξε υποστήριξη για το σχέδιο και μάλιστα ε, μας είπαν ότι έγιναν 125 συνεδριάσεις για να εγκριθούν τα υδρολογικά σχέδια με πάνω από 1.600 μέλη. 205 οργανώσεις συμμετείχαν. Υποβλήθηκαν 7.000 σχόλια στις συνεδριάσεις ή υπευλήθησαν και γραπτός. Ήταν τεράστια ε, η συμμετοχή και η διαβούλευση και ουσιαστικά τα υδρολογικά αυτά σχέδια, τα σχέδια διαχείριση λεκανών απορροή συγκέντρωσαν το 80% τη υποστήριξη όλων αυτών των πλατφορμών. Και επίση υπήρξε και το feedback τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έδωσε κάποιε κατευθυντήριε γραμμέ για τη βελτίωση κυρίω του δεύτερου κύκλου των σχεδίων διαχείριση και διαπιστώνω ότι αυτό το κάνει παραδοσιακά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υποβάλλει κάποιες συστάσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης. Το σημαντικό είναι να υπάρχει συνεργασία μεταξύ του τι λέμε εδώ, του τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της ανταπόκρισης που έχουμε από την Ισπανική κυβέρνηση. Νομίζω πάντως ότι πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Η Ισπανική κυβέρνηση στις, ε, στους δικούς της φορείς, γιατί έχουμε 13 ε, ε, οργανώσεις που εμπίπτουν στη τοπική αυτοδιοίκηση και 12 οργανώσεις και φορείς που εμπίπτουν στην κεντρική κυβέρνηση. Πάντως γίνεται συλλογική προσπάθεια για να τηρηθούν οι περιβαλλοντικές οδηγίες. Και από αυτή την άποψη και η κεντρική κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση τον ίδιο στόχο έχουν. Και όπω είπε η πρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν δεν υπάρξει μόρφωση με τι οδηγίε, θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Πάντω, αυτό που είπαμε στην έκθεση ε, τη διερευνητική αποστολή είναι ότι βρίσκεται σε σωστά χέρια η κατάσταση και η άγουσα είναι σωστή. Α περιμένουμε τις εκθέσεις Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να έχουμε το feedback τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πάντως έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στι ε, αρμόδιες αρχέ Και δεν μιλάω για συγκεκριμένη κυβέρνηση, γιατί οι κυβερνήσει πέφτουν ε, και οι τοπικές κυβερνήσεις επίσης αλλάζουν. Πάντως πιστεύω ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο με τη συλλογική προσπάθεια που έγινε στην Ισπανία και με τη συνεργασία και των κοινοτικών οργάνων. Η κυρία Ινέσα Γιάλα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρησή μου, γιατί δεν άκουσα από την αρχή ούτε τους ε, υποβάλλοντες την αναφορά ούτε ολόκληρη την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πάντως για τις πληροφορίες και την ενημέρωση. Εμένα με ενδιαφέρει κυρίως ο Εύρος γιατί είναι η γενέτειρά μου εκεί και γνωρίζω καλύτερα την περιοχή γύρω από τον Εύρο παρά την περιοχή γύρω από τον Τάγο. Πάντως εξασφαλίζουμε μια παρακολούθηση κατάστασης ε, μένουμε ενήμεροι και για τις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σίγουρα η λεκάνη απορροής του Εύρου είναι η πιο εκτεταμένη λεκάνη απορροής και είναι τόσο περίπλοκο το οικοσύστημα που χρήζει ιδιαίτερης φροντίδα και μέτρων. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε για τη σωστή διαχείριση. Επίσης, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στα ποτάμια αυτά, στα ποτάμια της Νότιας Ευρώπης, που έχουν ιδιαιτερότητες, γιατί είναι ποτάμια που έχουν διαφορετική μορφή το καλοκαίρι και το χειμώνα. Υπάρχει λειψιδρία, το καλοκαίρι ξεραίνονται τελείως. Υπάρχουν σχέδια στη μελλοντική διαχείριση ε, μέτρα θεκτικότητας και προσαρμογής κλιματικές αλλαγές. Γιατί ε, στον Εύρο το χειμώνα έχουμε τεράστιες πλημμύρες. Ευτυχώς φέτος δεν πλημμύρισαν τα χωριά, αλλά πλημμύρισαν τα χωράφια και χάθηκαν ολόκληρες οδιές λόγω και των ασταθών καιρικών συνθήκων φέτος. Οπότε υπευλήσαν πολλά αιτήματα για το καθαρισμό της Κίτης, του Εύρου, ε, που είναι περίπλοκα θέματα. Είναι σημαντικός ο διάλογος λοιπόν και με τους τοπικούς φορείς που είναι αρμόδιοι για τέτοιες ενέργειες. Και επίσης θα πρέπει να στηρίξουμε την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τις ε, ακολουθητές διαδικασίες για την εξασφάλιση του, του ύδατος σε, στο δέλτα του Εύρου, στις εκβολές. Επίσης, στην Αραγωνία έχουμε πρόβλημα με τους παραποτάμους του Εύρου. Και κάθε φορά συζητούμε την ανάγκη ε, της αντιμετώπισης ε, της ε, μόλυσης των εδαφών των παρόχθιων περιοχών. Μάλιστα, δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταφέρει να προωθήσουμε μια τέτοια οδηγία. Οδηγία ή κανονισμό. Τότε είχαμε προτείνει οδηγία για τα μολυσμένα εδάφη. Γιατί η ποιότητα του ύδατος, η ανθεκτικότητα, όλη αυτή η ικανότητα διαχείρισης του ύδατος που βρίσκεται στη λεκάνη απορροής σχετίζεται και με την ποιότητα των παρόχθιων εδαφών. Και αν είναι μολυσμένα αυτά τα ύδατα, ε, τα εδάφη θα μολυθεί και το είδωρ φυσικά. Και στην Ταραγώνα είχαμε ένα σχέδιο πιλωτικό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την μόλιση των παρόχθιων εδαφών. Ερωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι έγινε με την περίπτωση αυτή. Ίσως να μην είναι κατατοπισμένη η σημερινή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί κυρίως την ενδιαφέρει ε, η του ποταμού και μόλιση του ύδατος. Αλλά τότε είχαμε προτείνει μια οδηγία για τα μολυσμένα εδάφη, όχι μόνο για το είδωρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είναι σαφή η κατάσταση όπω διαμορφώνεται. Η σύσταση είναι να παραμείνει ανοιχτή εξέταση της αναφορά. Αλλά απευθύνθηκαν κάποιες ερωτήσεις προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω σοβαρότερο θα ήταν να μας αποστείλετε γραπτό τι απαντήσεις σας. Στείλτε δύο επιστολές. Μία για τις Ισπανικές Αρχές παρακαλούμε και μία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει των ερωτήσεών σα, για να λάβετε και μια επίσημη απάντηση γραπτή και θα συνεχίσουμε την εξέταση τη αναφορά. Ωραία. Πολύ ωραία. Και τώρα δύο λεπτά για, την, για τους αναφέροντες. Δύο λεπτά, όπως θέλετε να τα χωρίσετε εσείς μεταξύ σας. Oh, Αυτή τη φορά θα μιλήσω εγώ η Σουζάνα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που κρατήσατε ανοιχτή την αναφορά μας και δεν την αρχιοθετήσατε. Το πρόβλημα των υδρολογικών σχεδίων και της διαχείρισης των λεκανών απορροής είναι ένα θέμα που μας απασχολεί χρόνια ολόκληρα. Εξού και ο αριθμός των αναφορών που συστηματικά υποβάλλουμε και θα συνεχίσουμε, το φαντάζομαι στο μέλλον. Οι πολίτες νιώθουν μεγάλη απογοήτευση εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας είπε ότι το σχέδιο λεκανής απορροής ε, είναι αντικείμενο αγωγών και πολίτε έχουν προσφύγει στα δικαστήρια και είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι όσο εκκρεμωδικούν οι αποφάσεις δεν μπορεί να επέμβει. Εμείς ε, την ώρα που καταθέσαμε αγωγή στα δικαστήρια υποβάλαμε και την αναφορά ε, και γι' αυτό έχει κολλήσει το θέμα της αναφοράς περιμένοντας την απόφαση των δικαστηρίων. Δεν ξέρω αν φέτος την Άνοιξη ή το φθινόπωρο θα υπάρξει πρόοδος. Τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε τον προγραμματισμό του δεύτερου κύκλου. Αυτό που ζητήσαμε από την Επιτροπή, την αιτήση που υποβάλαμε στην Επιτροπή, δεν θα έχουμε χρόνο να την στηρίξουμε. Η Επιτροπή είπε ότι έκανε κάποιε στάσεις προ την Ισπανική κυβέρνηση που θα συμπεριληφθούν στο δεύτερο σχέδιο διαχείριση. Η πείρα όμω μα έχει δείξει ότι στην πράξη δεν λαμβάνονται υπόψη αυτέ οι στάσεις. Γιατί η συνομοσπονδία που εκπονεί τα σχέδια, παραλαμβάνω, δεν λαμβάνει υπόψη τις στάσεις Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Το είδαμε και στο πρώτο σχέδιο, οπότε νιώθουμε τελείως ανήμποροι. Είμαστε σαν ποντίκι, σαν χάμστερ που γυρίζουμε συνεχώ, προσπαθούμε να ανέβουμε σε αυτή τη ρόδα και δεν τα καταφέρνουμε. Πώς θα καταφέρουμε να συμπεριληφθούν αυτές οι τάσεις, να ληφθούν υπόψη και να εφαρμοστούν από την Ισπανική κυβέρνηση, γιατί δεν υπάρχει αλλαγή στην οτροπία σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό. Δυστυχώς ε, το νερό αντιμετωπίζεται ως ε, οικονομικό εμπορεύσιμο αγαθό και ξεχνούν ε, πολλοί ότι το είδωρο δεν έχει μόνο οικονομική, αλλά και περιβαλλοντική και οικολογική αξία. Πριν από δύο εβδομάδες ε, ε, γιορτάσαμε τους υγρότοπους στην Ισπανία και δώσαμε έμφαση στο δέλτα του Εύρου. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η υποχώρηση των υδάτων λόγω της ε, κατακράτησης των ειζημάτων στα φράγματα. Μάλιστα του χρόνου, το συγκεκριμένο σημείο του Εύρου στο οποίο ε, είχαμε τις εκδηλώσεις δεν θα υπάρχει. Γιατί γίνεται τέτοια υποχώρηση ε, που σε μερικά σημεία είναι 4 μέτρα, σε άλλα 16 μέτρα. Φανταστείτε, φέτος βάζετε την πετσέτα σε ένα σημείο ε, το, της όχθης και του χρόνου δεν θα υπάρχει αυτό το σημείο. Αυτό το πρόβλημα έχουμε με το Δέλτα του Εύρου, γιατί η διαχείριση της λεκάνης απορρίσης του Εύρου δεν λαμβάνει υπόψη ε, την κατάσταση κατάντη. Μπορεί να ξεπέρασα το δίλεπτο και σας ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, αλλά έπρεπε να τα πω. Ο κύριος Αγγιλάρ. Ευχαριστώ καταρχήν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την, την Επιτροπή σας μάλλον, την Επιτροπή Αναφορών που κράτησε ανοιχτή την αναφορά. Και όπως είπε η κυρία Μποντήλ Βαλέρο, ο τάγος έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά και σχεδόν δεν υπάρχει ελπίδα για την ανάκτησή του, γιατί για να ανακτήσουμε την κατάσταση του τάγου, του τάγου θα πρέπει τα περιβαλλοντικά συμφέροντα να υπερισχύσουν των οικονομικών. Επίσης, ε, αυτά τα μερκαντιλιστικά συμφέροντα, όπως είπα, δεν είναι βιώσιμα, γιατί ουσιαστικά θέλουμε να σφάξουμε την κότα που κάνει το χρυσό αυγό. Ε, δυστυχώς, ε, η εκτροπή του σεγούρα προς τον, προς τον ε, τάγο συνεχίζεται, κάτι που επιδεινώνει την κατάσταση. Η κατάσταση στην Ανατολική Ισπανία είναι μη βιώσιμη. Θα εξαφανιστούν τελείως τα ποτάμια μας. Περιμένουμε την έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα μας πει όμως αυτό που γνωρίζουμε ήδη. Η Ισπανική κυβέρνηση και οι Ισπανικοί φορεί δεν συμμορφώθηκαν με τις υποχρεώσεις της οδηγίας πλαίσιο για το είδωρ και διαπιστώσετε κι εσείς με τα μάτια σας την κατάσταση στα δύο ποτάμια. Δεν προσπαθούμε να σας πείσουμε γιατί το είδατε και με τα μάτια σας και έχετε νομίζω πιστεί θα πρέπει να εφαρμοστεί κοινοτική νομοθεσία. Δεν ζητήσαμε τίποτα καινούριο, ούτε τίποτα φοβερό. Ζητήσαμε απλώς ότι θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις της οδηγίας πλαίσιο για το είδωρ. Θα πρέπει να τηρηθούν οι, δια... διατάξεις αυτές και για τον τάγο, που είναι περιβαλλοντική αρτήρια της κεντρικής Ισπανίας. Καταστρατηγείται όχι μόνο η οδηγία πλαίσιο για το είδωρ, αλλά και άλλες περιβαλλοντικές οδηγίες. Θα πρέπει να φέρουμε την Ισπανική κυβέρνηση και τις Ισπανικές αρχές ενώπιον των ευθυνών τους. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τα δικαστήρια να αποφασίσουν για όλες τις αγωγές. Σε κάθε εκτροπή που γίνεται υποβάλλεται διοικητική αγωγή. Κάθε μήνα έχουμε τέτοιες αγωγές. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να ε, διευθετηθούν όλες αυτές οι αγωγές είτε σε διοικητικά δικαστήρια είτε αλλού γιατί θα φτάσουμε σε σημείο χωρίς επιστροφή, σε μια κατάσταση μια αντιστρέψιμη. Οπότε θα πρέπει να μην μείνει ανοιχτή αναφορά όπως είπατε, αλλά θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί αν δεν ξεκίνησε ήδη η διαδικασία επιπαραβάση κατά τη Ισπανική κυβέρνηση, πότε θα το κάνει. Θα πρέπει επιτέλους να τηρηθεί η οδηγία πλαίσια για το είδωρο. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώνουμε τώρα με αυτές τις αναφορές το επόμενο θέμα είναι η επίσκεψή μας στην Σλοβακία ορίστε ναι ναι βεβαίως Γενικά θα είναι καλύτερα γραπτός, αλλά μπορείτε να μας τα πείτε κιόλας. Ευχαριστώ, θα είμαι επιγραμματική. Περιμένουμε τις παρατηρήσεις ε, και γραπτός. Θα ήθελα πάντως να τονίσω και πάλι ότι επίκειται η δημοσίευση ενός πακέτου εκθέσεων που αφορά τη διαχείριση ε, των λεκανών απορροής και την τήρηση της οδηγίας πλαίσια για το είδωρ. ονούπο θα δημοσιευθούν οι σχετικές εκθέσεις θα έχετε πιο σαφή στοιχεία. Άλλωστε, στις εκθέσεις αυτές έχουμε πολύ συγκεκριμένα θέματα. Την υποχρέωση για τις οικολογικές ροές, τις εξε, εξαιρέσεις και το θέμα της ανάκτησης του κόστους. Αυτά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε λοιπόν με την επίσκεψή μας στην Σλοβακία. Και βεβαίω ε, υπάρχει έτοιμο να μιλήσουμε και για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Ο επικεφαλή αντιπροσωπεία ήταν η κυρία Σεσίλια Βίξτρομ. Μα ζητάει να αποστείλουμε λοιπόν τρει επιστολέ στο κάθε κράτος και να ζητήσουμε περισσότερε πληροφορίε για την τρέχουσα κατάσταση τώρα θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Μπιαλκοβίτσοβα, από την DJ Η Κομισιόν ακολούθησε την σύσταση που λάβαμε. Σημειώσαμε τις συστάσεις, ήρθαμε και σε επαφή με την ε, Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για να δούμε τα ζητήματα αυτά. Η Κομισιόν λοιπόν παρακολουθεί την κατάσταση στην Σλοβακία και στην Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Τα έχουμε καταγράψει αυτά όλα και η επόμενη έκθεση θα δημοσιευτεί σε μία εβδομάδα και θα υπάρξει και ο κατάλογος των επενδυτικών προτεραιοτήτων του ΕΣΥΦ Οπότε παρακολουθούμε τις προτάσεις αυτές ε, και τις ανάγκες που υπάρχουν. Επίσης επενδύουμε την διαδικασία αυτή ήδη από τώρα υπάρχουν επενδύσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το ΕΚΤΠΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο επικεντρώνεται περισσότερο στην ε, κατάρτιση ενώ βεβαίως το ΕΚΤΠΕ ε, στις υποδομές ε, έχουμε βεβαίως και κάποιους όρους εξάντε άντε αιρεσιμότητα ειδικά όσον αφορά την διοικητική ικανότητα για την εφαρμογή της σύμβασης ε, του ΟΗΕ για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία. Οπότε... Σημειώνουμε πλήρως τις συστάσεις της έκθεσης, ε, ειδικά στα θέματα των όσων έχουν εφαρμόσει τα κράτη-μέλη σύμφωνα με το πρόγραμμα. Στη Σλοβακία μπορώ να σας πω ότι Μέχρι στιγμής είχαμε έξι γύρους διαγωνιστικής διαδικασίας ε, για επενδύσεις 67,4 εκατομμυρίων και αναμένονται να υπάρξουν και άλλες προκηρύξεις διαγωνισμών για να έχουμε και άλλες ε, επενδύσεις σε υποδομές. Υπάρχει λοιπόν ένα σαφής ορισμός του τι θέλουμε να υπάρξει Υπάρχει το όριο των 12 ατόμων σε ένα κτίριο, όμως ε, εδώ πέρα η Σλοβακική Υπηρεσία θέλει να βάλει 40 άτομα σε ένα κτίριο και έχουμε άρα κάποιες ε, δυσκολίες στην εφαρμογή αυτών των μέτρων γιατί δεν θέλουν ε, και οι δικαιούχοι να ακολουθήσουν αυτόν τον περιοριστικό ορισμό αυτό μπορώ να πω αυτήν την ε, στιγμή για την έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποιος άλλος. Όχι, κοιτάξτε, και εγώ Σλοβάκος ε, είμαι, Σλοβάκος πολίτης. Ε, ξεκάθαρα τα πράγματα, αλλά Υπάρχουν και κάποιες περιπλοκέ. Θα ήθελα λοιπόν να επαναλάβω το αίτημα τη κυρία Βίξτρομ να αποσταλούν οι επιστολέ αυτές για περαιτέρω πληροφορίε. Τι είναι? Τρεις επιστολέ μόνο για πληροφορίε, μάλιστα. Το επόμενο θέμα αφορά την επίσκεψή μας στην Σουηδία. με βάση το αίτημα του ΕΛΚ και των φιλελευθέρων ήμουν και εκεί επικεφαλής της αντιπροσωπείας και υπήρχαν κάποια σοβαρά προβλήματα στην Σουηδία. που αφορούσε το ζήτημα του αριθμού ταυτότητας ε, πολιτών της Ένωσης. Και πάλι λοιπόν υπάρχει εδώ πέρα η θέση της κυρίας Βίξτρομ. Οπότε θα ήθελα να ακούσουμε τους ε, αναφέροντες ε, ποιος είναι εδώ ο κύριος Άντωνη Βάλκε. Έχετε τον λόγο για 5 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ που μας ε, καλέσατε στην ε, σημερινή ακρόαση για το θέμα αυτό. Άντωνι Βάλκ είμαι από μια οργάνωση για τα ευρωπαϊκά δικαιώματα και ένα συνάδελφος από το Crossroads Göteborg. Όπως ξέρετε, το θέμα αυτό κρατάει σχεδόν 10 χρόνια. Η πρώτη ε, αναφορά που λάβατε είναι από το 2010. Το πρόβλημα είναι ότι οι Σουηδικές αρχές αρνούνται να εκδώσουν αριθμό αφημί σε Ευρωπαίους πολίτες που κατοικούν νόμιμα στη χώρα. και διάφοροι πολίτες που σπουδάζουν ή έχουν κάποια βραχυπρόθεσμα Κάθε βραχυπρόθεσμες συμβάσεις ε, δυστυχώς ε, δεν καταγράφονται από τις φορολογικές αρχές. Γιατί είναι πρόβλημα αυτό. Γιατί οποιοδήποτε ζει στην Σουηδία χρειάζεται τέτοιον αριθμό για να έχει πρόσβαση και σε άλλες ε, δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες. Αυτό το έχει επιβεβαιώσει και το εμπορικό επιμελητήριο της Σουηδίας που επιβεβαιώνει ότι όλες σχεδόν οι υπηρεσίες πλέον στην Σουηδία σχετίζονται με τον προσωπικό αυτόν αριθμό. Οπότε χρειάζεται αυτός ο αριθμός. Και προφανώς πολλές από αυτές οι υπηρεσίες έχουν ψηφιοποιηθεί και το πρόβλημα γεροτερεύει για όσους ε, δεν έχουν ε, προσωπικό αριθμό. Χωρίς λοιπόν προσωπικό αριθμό ε, δεν μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση. Δηλαδή μιλάμε για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού. Συστημένα δέματα για να παραλάβει για να παρακολουθήσει μαθήματα σου ειδικής γλώσσας δωρεάν, για πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας ε, και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι μακρύς ο κατάλογος των υπηρεσιών που πλέον απαιτούν ε, προσωπικό αριθμό και χωρίς αυτόν δεν υπάρχει πρόσβαση. Το πρόβλημα λοιπόν πηγάζει από τους κανόνες περί καταγραφής στο ε, ληξιαρχείο σύμφωνα με τους κανόνες περί ε, λήξη αρχείου, το άρθρο 3 συγκεκριμένα, μόνοι όσοι μπορούν να ε, επιδείξουν ότι θέλουν να παραμείνουν στη Σουηδία για πάνω από ένα χρόνο, μπορούν να εγγραφούν στο λεξιαρχείο. Και θεωρείται κάποιος κάτοικος όταν θα περνάει ε, τον ελεύθερο χρόνο του στη χώρα τουλάχιστον για ένα έτος. Τι σημαίνει ελεύθερος χρόνος? σημαίνει ότι όταν ε, δεν εργάζονται σε καθημερινή ή σε εβδομαδιαία βάση θα κάθονται στη Σουηδία. Δηλαδή βασικά ο νόμος ε, έχει σχεδιαστεί για άτομα που θα παραμένουν για πάνω από ένα έτος. Το πρόβλημα είναι η πρακτική εφαρμογή ε, των κανόνων ε, από τις ε, φορολογικές αρχές που κάνουν μια πολύ περιοριστική ερμηνεία για να μπορούν οι άνθρωποι να αποδείξουν ότι κατοικούν στη Σουηδία πάνω από ένα χρόνο. Το πρόβλημα είναι βεβαίως ότι οι πολίτες της Ένωσης δεν έχουν αυτό το προνόμιο εάν έχουν βραχυπρόθεσμα συμβόλαια ή ακόμα και αν ζουν σου ίδια πάνω από ένα χρόνο απορρίπτονται. Λοιπόν, ο χρόνος ε, τελειώνει. Θα αναφερθώ ε, σε κάποιες από τις συμβαστικές προτάσεις ε, της Σουηδικής κυβέρνησης. Το κράτος προτείνει να επεκταθεί η χρήση του προσωπικού αριθμού. Δεν είναι λύση αυτό. Δεν, του αριθμού συντονισμού, όπως λέγεται. Μα δεν υπάρχει παροχή στις πρόσβαση με συγχωρείτε στις υπηρεσίες ε, και αυτός ο αριθμός επίσης ε, δίνεται σε άτομα που μπορούν να αποδείξουν διαμονή 6 μηνών. Και εκεί πέρα λοιπόν προκύπτουν προβλήματα. Και πολλοί από τους ιδιωτικούς πάροχους υπηρεσιών δεν αναγνωρίζουν τον αριθμό συντονισμού. Γιατί? γιατί ο προσωπικός αριθμός βασίζεται στην ημερομηνία γέννησης. Ο αριθμός συντονισμού έχει την ίδια προσέγγιση, αλλά προσθέτει ε, το 60 στην ημερομηνία γέννησης. Οπότε τα συστήματα πληροφορικής δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τον αριθμό συντονισμού. Οπότε η πρόταση της Σουηδικής κυβέρνησης απλά θα δημιουργήσει κόστος στις επιχειρήσεις. Ποιος θα το πληρώσει αυτό. Οι επιχειρήσεις δεν θα αλλάξουν τα συστήματά τους ε, επειδή τους το λέει το κράτος. Οπότε, δυστυχώς δεν είναι λύση αυτό. Ζητάμε λοιπόν από την Επιτροπή σας να αναλάβει δράση. Πρώτον, η Σουηδική κυβέρνηση αναφέρεται σε κάποιες εκθέσεις ε, τις οποίες δεν μας τις δίνει. Μετά η απάντηση της κυβέρνησης μας δείχνει πως οι κανόνες των εφοριακών αρχών έχουν αλλάξει. Αλλά δεν μας λέει ποιες είναι αυτές οι αλλαγές. Είδαμε τις νέες κατευθυντήριες γραμμές. Δεν βλέπουμε κάποια ουσιαστική αλλαγή. Δυστυχώς. Όλες οι δράσεις μας λέει ότι έλαβε το Σουηδικό κράτος δεν έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Οπότε ζητάμε να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή και να κανονίσουμε κάποια στιγμή αργότερα μια ακρόαση για να δούμε τις εξελίξεις όταν μας δώσει τις μελέτες ε, στις οποίες παραπέμπει το Σουηδικό κράτος. Με συγχωρείτε που ε, μακρηγόρησα, αλλά είναι σημαντικό το ζήτημα και ελπίζω να κρατήσετε την αναφορά ανοιχτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα τώρα να ακούσουμε την κυρία Μόνικα Μούσα από την Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλή μέρα σας. Συμφωνούμε τις ανησυχίες του κυρίου Βάλκε Γι' αυτό ακριβώς είμαστε σε επαφή με τις Ιουδικές Αρχές εδώ και χρόνια και μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ο Γενικός Διευθυντής συναντήθηκε με τις ειδικέ Αρχές για να δούμε το πού βρισκόμαστε. Το πρόβλημα με τον αριθμό αυτών είναι διτό. Λάβαμε κάποιες καταγγελίες για το ότι κάποιος ο οποίος δεν έχει οικονομική δραστηριότητα δεν μπορεί να έχει ιδιωτική ασφάλιση υγείας η οποία θα αναγνωρίζεται ως τέτοια υπήρχε πρόβλημα στο να λάβει τον αριθμό αυτόν, αλλά αυτό μάλλον λύθηκε με τις περσινές κατευθυντήριες γραμμές. Τώρα αποδέχονται την ασφάλιση υγείας στις Σουηδικές Αρχές, οπότε ελπίζουμε να μην υπάρχουν άλλες τέτοιες δυσκολίες. Βεβαίως το πρόβλημα παραμένει ε, δεν μπορούν δηλαδή τα άτομα να λάβουν ε, προσωπικό αριθμό αν δεν παραμείνουν για πάνω από ένα έτος. Η Κομισιόν ζήτησε από τις Σουηδικές Αρχές να αναζητήσουν λύσεις να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες αυτές και πράγματι ε, μία από τις απαντήσεις είναι η χρήση του αριθμού συντονισμού ο αριθμός συντονισμού στο μέλλον ε, μας είπαν οι Σουηδικές Αρχές ε, ότι θα νομοθετήσουν ώστε να καταστεί πιο χρήσιμος για να μπορούν οι άνθρωποι να ζητάνε τέτοιον αριθμό. Επίσης ε, θέλουν να γίνει ο αριθμός πιο αξιόπιστος και βεβαίως οι αρχές γνωρίζουν την ταυτότητα του ετούντος για να μπορούν να δεχτούν τον αριθμό και οι αρχές και οι ιδιώτες. Επίσης, οι Σουηδικές Αρχές θα κάνουν μια εκστρατεία ενημέρωσης και βεβαίως με τα μέτρα αυτά τα άτομα τα οποία έχουν ένα αριθμό συντονισμού θα μπορούν να ζουν όπως ε, και τα άτομα τα οποία θα έχουν ε, προσωπικό αριθμό. Βεβαίω δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι έχουν να μας πούν κάτι. Παρακαλώ. Απλώς να παρέμβω και να πω ότι βάσει των όσων είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η σημαντικότατη αυτή αναφορά που συζητούμε και ήταν και αντικείμενο διερευνητική αποστολή. Είναι μια αναφορά που πρέπει να συνεχίσει να εξετάζεται και ελπίζω η συμφωνία να εφαρμοστεί στο δυνατόν γρηγορότερα για να επιληθεί το πρόβλημα αυτό που είναι πολύ ε, λεπτό για τους αναφέροντες. Πρόεδρος αυτό που ζητάτε είναι ακριβώς ε, το ίδιο με αυτό που ζητάει και η υπόλοιπη Επιτροπή Αναφορών και η Πρόεδρος και του Προεδρείου. Θα φροντίσουμε να αποδεθύνουμε επιστολή στη Σουηδική Κυβέρνηση. Και τώρα ο κύριος Βάκελ, ο κύριος Βιτόρια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, εκτιμούμε τις προσπάθειες που καταβάλει η Επιτροπή Αναφορών σας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προσπαθήσουν να βρουν μια λύση στο πρόβλημα του προσωπικού αριθμού. Το βασικό πρόβλημα είναι τα προβλήματα της Σουηδικής κυβέρνησης και πώς θα μεταφραστούν σε ε, πράξη. Εάν ο αριθμός συντονισμού είναι μια λύση ενδιάμεση, θα χρειαστεί νομοθεσία για να καταγραφεί αυτό. Θα χρειαστεί νομοθεσία για να είναι υποχρεωτική η χρήση του και να μπορεί κανείς να επιτρέψει στους συγγενείς και τα μέλη της οικογένειας να έχουν πρόσβαση ακριβώς στις ίδιες υπηρεσίες. Το θέμα που αναφέρθηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες είναι ένα θέμα ε, για το οποίο λαμβάνουμε ακόμη προσφυγές ε, προσφυγές από κόσμο που δεν λαμβάνει αγωγή υπερήθαλψη ε, γιατί δεν έχει περσό number. Ε, πρέπει λοιπόν η ειδική κυβέρνηση να αναλάβει τις δεσμεύσεις αυτές κάποια στιγμή να τις ε, τηρήσει και να κάνει κάποια αλλαγή στην πράξη. Ε, παρακαλούμε να συνεχίσετε να παρακολουθείτε το θέμα και εσείς Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να δώσω λίγο το λόγο και στο συμβάλιο, το, το, συγγνώμη, στο συνάδελφο, τον Φαμπρίτσο Βιτόρια, γιατί δεν τον άφησα να μιλήσω τώρα. Καλημέρα σε όλους. Το πρόβλημα με τον αριθμό συντονισμού είναι ότι δίνεται σε ανθρώπους που έχουν μείνει λιγότερο από ένα χρόνο στη Σουηδία. Κάτι που είναι παραβίαση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την Ελευθερία της Κυκλοφορίας του 2008 εδώ γίνεται διάκριση μεταξύ ανθρώπων που μένουν ε, λιγότερο από έναν χρόνο με αυτούς που μένουν παραπάνω. Δεν υπάρχει καμία διάταξη στην Ευρωπαϊκή Οδηγία ή στην ε, σχετική νομοθετική πράξη τη Σουηδία που τη μεταφέρει που να χωρίζει τους κατοίκου σε δύο κατηγορίες. Ευρωπαίου πολίτε δηλαδή που έχουν μείνει λιγότερο από περισσότερο από ένα χρόνο. Υπάρχει εδώ ένα θέμα ε, αντικειμενικότητας. Δεν μπορεί να γίνεται διαχωρισμό. Ο κόσμο έχει φύγει από τη Σουηδία, έχει εκπληρώσει τι προποθέσει τη Ευρωπαϊκή Οδηγία. Πρέπει να αναγνωρίζεται ω ε, διαμένον, ω κάτοικο, με τον ίδιο τρόπο που αναγνωρίζονται οι Σουηδοί πολίτε. Το να γίνεται τέτοια διαφοροποίηση με τον αριθμό συντονισμού και όχι με το περσό number, ε, είναι διακριτική μεταχείριση βάσει των δικαιωμάτων ελεύθερη κυκλοφορία. Ευχαριστούμε πολύ για τους δύο αναφέροντες και τώρα πάμε στην Ιταλική αναφορά. Υποδέχομαι εδώ τους κυρίους, τις κυρίες Πίβα, τον κύριο Μαντοβάνη και τον κύριο Τσινέζη που είναι οι αναφέροντες, είναι παρόμοιες μεταξύ τους οι αναφορές. Θα δώσω το λόγο στην Μικαέλα Πίβα για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Πρόεδρε. Εδώ έχουμε έρθει για την αναφορά για την ε, επέκταση της εμπορική, του εμπορικού κέντρου στο Αρέζε. Μια επέκταση μαζικότατη για την έκταση μιας βιομηχανικής περιοχής της Αλφα Δηλαδή αυτή η περιοχή που αρχικά τη χρησιμοποιούσε η για παραγωγή τώρα θα γίνει ουσιαστικά ένα εμπορικό κέντρο. Το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο τη Ευρώπης είναι ο στόχος. Και θα διπλασιαστεί η έκταση των εμπορικών ε, χώρων. Δεν βλέπω τις διαφάνειες όμως. Α, ωραία. Σε κάθε περίπτωση το πολεοδομικό σχέδιο θα επηρεάσει την ε, κίνηση, την ατμοσφαιρική ρήπανση, την ποιότητα δηλαδή του αέρα και το πώς θα λειτουργούν τα εμπορικά καταστήματα που δεν θα υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτούς που ίσχυαν και εγκρίθηκαν πρόσφατα. Το πρόβλημα είναι λοιπόν οι περιβαλλοντικοί δείκτες που θα, θα χειροτερέψουν και θα επηρεαστεί η υγεία των πολιτών. Το πρόγραμμα, όλο έργο, να και Και βλέπουμε και την φωτογραφία αεροπλάνο που ε, προβλέπει από 7.500 τετραγωνικά μέτρα να περάσουμε σε 150.000 τετραγωνικά μέτρα. Αυτή είναι η τελική μορφή της επέκτασης. Βλέπετε το, ε, το σχέδιο το 2016 δεν έχει αλλάξει και το πρόβλημα είναι ότι οι τρεις δήμαρχοι των δήμων που ε, είναι όμοροι αυτής της περιοχής συζητάνε για το όλο πρόβλημα. Η ε, αγορά του Σιντόρ ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί θα υπάρχουν ε, σίγουρα μια μεγάλη ανοιχτή περιοχή, κάποιο είδους μέγαρο, δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί τι μορφή θα έχει. Και έχουμε καταφέρει να πάρουμε εκτιμήσεις για το πώς θα θα διαμορφωθεί κίνηση των αυτοκινήτων. 43.000 οχήματα και 2.300 είναι ε, στις ώρες εχμής η κίνηση των οχημάτων. Τώρα με την... Τώρα με τη νέα ε, οδό που θα δημιουργηθεί θα, υπάρχει 46, θα υπάρχουν θα υπάρξουν 46.070 οχήματα, διπλασιασμός πλήρης δηλαδή και μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στην πλέον ε, μολυσμένη περιοχή της Ευρώπης από την πλευρά της ατμοσφαιρικής ρήπανσης, στην κοιλάδα του Πάδου ε, στην ε, Ευρώπη. Ε, το θέμα της οδηγίας λοιπόν για την ατμοσφαιρική ρήπανση είναι κέριο εδώ, διότι μιλάμε για την μόλυνση που προκαλούν τα οχήματα. Και θα έχουμε 100% αύξηση της κίνησης σε σχέση με την τωρινή προβλέπονται 15.000 περισσότερε θέσει αυτοκινήτων. Ε, έχουμε επισημάνει τα στοιχεία αυτά από το 2016 βάσει τις οδηγίες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Έχουμε συγκεντρώσει επί σειρά ημερών τις τιμές των ε, ρήπων στον, ε, στην ατμόσφαιρα το 2017. Τα αποστήλαμε και τα επεξεργάστηκε η ο τοπικός φορέα του Αρέζα για το περιβάλλον, η ε, κάποια τον Αύγουστο του 2018, το γραφείο αυτό έκλεισε. Δεν έχουμε πλέον άλλα δεδομένα συγκρίσιμα να σας δώσουμε πιο πρόσφατα το γραφείο για την προστασία του περιβάλλοντος δεν έχει λειτουργήσει εδώ και σε 147 ημέρες. Άρα από τα στατιστικά δεδομένα, από τους πλέον μολυσμένους δήμους στην ε, περιοχή του Μιλάνου από το 2016-2018, έχουμε φτάσει να είμαστε λιγότερο. Διότι έχουν κατέβει τα δεδομένα μας σε σχέση με το μέσο όρο, αλλά δεν έχει αλλάξει τίποτα σε τοπικό επίπεδο. Είμαστε ε, ένας δήμος που μα κλείνει από δύο πλευρές, κλείνουν από δύο πλευρέ δύο αυτοκινητόδρομοι που οδηγούν προ άλλε πόλει από το Μιλάνο. Οπότε είναι τεράστια η κυκλοφορία οχημάτων. Ω προ το κέντρο, οι συμφωνίε και τα συμβόλαια έκλεισαν πριν από λίγο καιρό. Η ΑΡΠΑ έχει αναλάβει την ε, εκτέλεση, ΑΡΠΑΚ μάλλον, η οποία συγκεντρώνει τα δεδομένα και οι τα περιβαλλοντικά στοιχεία συγκεντρώνονται, με, έχουν ζητηθεί από την εταιρεία, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα. Ε, τι γίνεται λοιπόν με όσα έχουμε συγκεντρώσει. Θα πρέπει να υπήρχε ένας ιστότοπος ο οποίος να ε, ενημερώνεται με τα περιβαλλοντικά δεδομένα. Δεν υπήρχε. Εμείς λοιπόν φροντίσαμε να τα πάρουμε από το περιβαλλοντικό περιτηρητήριο της περιφέρειας της Λομβαρδίας. Και δεν υπάρχει άλλη... Ε, δεν έχει δοθεί καμία προθεσμία ως προς τα δεδομένα για την υγεία του πληθυσμού που θα έπρεπε να συγκεντρώσει ο τοπικό φορέας για την προστασία τη υγείας των πολιτών έχουμε παρατηρήσει αύξηση στην περιοχή του Αρέζε ε, όγκων, όγκων ε, θανάτων μάλλον λόγω όγκων. αυτό δεν είναι βέβαια σαφέ, διότι δεν έχουμε όλου του θανάτου καταγεγραμμένου στο ληξιαρχείο. Υπάρχει αύξηση 200% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τελευταία τριετία. Κοιτάξαμε και τα στοιχεία για τι καρδιοαγγειακές παθήσεις που έχουν αυξηθεί κατά 150%. Όλα αυτά τα στοιχεία τα έχει δει και ο τύπος, έχουν προσελκύσει την προσοχή των δημοσιογράφων ε, και για την ώρα τα δεδομένα που έχουμε, παρόλο που δεν είναι πάντοτε πρόσφατα, είναι πολύ ανησυχητικά, ιδίω αυτά περί της υγείας. Για τις χρόνιες καρδιοαγκιακέ παθήσεις έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην καταγραφή τους από τον τοπικό φορέα. Δεν ξέρουμε γιατί. Ε, η περιφέρεια τη Λομπαρδία και ο Δήμο του Μιλάνου ξεπερνάει το μέσο όρο, ιδίω για τι καρδιοαγγειακές Και σε σχέση με τη βιώσιμη κυκλοφορία, να σα ζητήσω να μιλάτε λίγο σιγά. Σιγά λόγω της μετάφρασης. Ναι, τα πρωτόκολλα για την ατμοσφαιρική ρήπανση είναι σημαντικά, ε, αλλά εάν οι εταιρείε εκεί βασίσουν ε, τα κέρδη τους στην κίνηση των οχημάτων, δεν θα γίνει τίποτα για τις παθήσεις. Τι να πούμε για τη βιώσιμη δηλαδή κινητικότητα, αν δεν λάβουμε υπόψη και τις επιπτώσεις στην υγεία. Ε, επιπτώσεις οι οποίες στη δική μας την περιοχή πολλαπλασιάζονται. Έρχεται σε αντιδιαστολή αυτό με την οδηγία για τον ατμοσφαιρικό αέρα η βιώσιμη ανάπτυξη δυσκολεύεται σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Θα θέλαμε λοιπόν να γίνει κάτι και να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς αυτής. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο λόγος στον Μασιμιλιάνο Μαντοβάνη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε αυτό το θέμα σήμερα. Προσπαθήσαμε και σε διάφορες, σε άλλα θεσμικά επίπεδα να ακουστεί το αίτημα μας, όμως τώρα Αυτή η περίπτωση που θα σα παρουσιάσουμε είναι μια εμπορική δραστηριότητα που συνεχίζει να ενόχληται χωρί καμία αντίσταση προ την προς τη Για τη δική μα την αναφορά σε σχέση με την προηγούμενη και την επόμενη, Υπάρχει το πρόβλημα των δυσκολιών που θα δημιουργήσει στον Πολάτε ένα καινούριο εμπορικό κέντρο. Πάλι πάντα στην περιφέρεια του Μιλάνου, στη, στα βόρεια της πόλης. Θα συγκεντρωθούμε σε δύο πτυχές. Πρώτα απ' όλα τη ρήπανση. Ακούσαμε και από την προηγούμενη αναφορά ποια είναι τα προβλήματα. Έχουμε προβλέψει κάποιες διαφάνειες Διότι γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρόλα, παρόλο που γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει πολύ καλά την ε, κατάσταση τη ρήπανση σε όλη μα την ε, περιοχή, τη γεωγραφική αυτή περιοχή και την κοιλάδα του Πάδου. Η διαφάνεια αυτή προσπαθεί να παρουσιάσει την επικράτεια που συζητάμε. Έχουμε μία επικράτεια πολύ μολυσμένη που κάνει πολύ λίγα για να μειώσει την ρήπανση αυτή. Ε, έχουν επιβληθεί και κυρώσεις στην Ιταλία για αυτόν τον λόγο, ιδίως στην ε, περιοχή της Λομπαρδίας. Ακούσαμε ότι αυτό που ακριβώς συμβαίνει είναι ότι τα γραφεία αυτά, οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή των στοιχείων, κλείνουν. Και τα έργα προχωρούν ανενόχλητα. Βλέπετε εδώ μια διαφάνεια που παρουσιάζει με κόκκινο μια περιοχή όπου κατά κύριο λόγο φαίνεται πόση ρήπανση υπάρχει από άζωτο, από ρήπους που επηρεάζουν ιδιαίτερα την υγεία. Και εδώ βλέπετε με το κόκκινο κυκλάκι που βρίσκεται η ρήπανση του μικροσωματιδίου 10, ιδίως ε, για τις περιοχέ με το κόκκινο κυκλάκι ισχύει αυτό, αλλά είναι όλη η περιφέρεια της Λομβαρδία από το 2016. Η κατάσταση δεν έχει αλλάξει πολύ εκ τότε. Εδώ βλέπουμε το διοξίδιο του αζότου, το διοξίδιο του αζότου, μια κατάσταση πολύ ανησυχητική. Και αυτός είναι ένας πίνακας, ο οποίος Μα ε, μας έχει έρθει από την ίδια την εταιρεία που θέλει να χτίσει το εμπειρικό κέντρο. ένα πίνακα που δείχνει ξεκάθαρα πώς θα αυξηθεί η κίνηση των αυτοκινήτων, η κίνηση οχημάτων, μάλλον πώς θα επηρεαστούν τα διάφορα αέρια, οι ρήποι που εκλείονται, αυτοί που είναι πλέον μολυσματικοί και η πιο βλαβερή για την υγεία. Η ρήπανση και οι συνέπειες στην υγεία. Δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε εμεί ποιε είναι οι ζημιέ για την ανθρώπινη υγεία. Υπάρχουν μελέτε που το αποδεικνύουν. Ε, τα μικροσωματίδια αυξάνει τι περιπτώσεις ε, φλεγμόνων και λοιμόξεων ε, αναπνευστικών και των ε, όγκων. Είναι κάτι ανάλογο και για την Εθάλη. Ε, αυτά τα στοιχεία έρχονται από, το Ευρωπαϊκό, από την τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για το Περιβάλλον και δείχνουν πόσο ανησυχητικά είναι τα πράγματα στην περιοχή μας. 35 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες ζουν σε ιδιαίτερα μολυσμένες περιοχές. 3,7 εκατομμύρια είναι οι και μόνο της κοιλάδας του Πάδου. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο τοποθετούμαστε. Για να μην εξηγήσω τώρα τα υπόλοιπα έργα για τα οποία έχουμε υποβάλει αναφορά, ε, είναι υποδομές. Ε, το πραγματικό όμως πρόβλημα, πρόεδρε και βουλευτές, δεν είναι το ίδιο το έργο είναι το σύνολο των έργων που θα εκτελεστούν και το σύνολο των υποδομών που δημιουργούνται στην περιοχή αυτή. Υπάρχουν σοβαρότατες αυξήσει. Ακούσαμε πλήν στο Αρέζε το 100%, εμείς είμαστε στο 20% περίπου της αύξησης της ρήπανση. αλλά γίνονται όλα ταυτόχρονα. Και ενώ ο στόχος μας είναι να καταπολεμήσουμε τη ρήπανση, εδώ δείχνουμε ότι θα αυξηθεί πολύ και πολύ γρήγορα μερικά στοιχεία και για την ε, καταστροφή, τη φθορά του εδάφους. Διότι στην περίπτωσή μας, όπως θα δείτε και στη διαφάνεια, μιλάμε για αυτήν ακριβώς την περιοχή. Είναι μια περιοχή τελείως αγροτική, αγροτεμάχια είναι, τα οποία σε επίπεδο πολεμπομίας έχουν καταγραφεί τα αγροτεμάχια ως εμπορική ζώνη, αλλά υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ του τι λέει το κτηματολόγιο ε, και το τι πραγματικά συμβαίνει. Εάν δείτε την φωτογραφία, πού είναι το εμπορικό στην ε, συγκεκριμένη περιοχή. Είναι ένα πράσινο λιβάδι. Ένα αγροτεμάχιο που θα μπορούσε μάλιστα να λειτουργήσει σαν αντισταθμιστικός παράγοντας για τη μόλυνση που έχουμε για τα νερά στην επιφάνεια, για τους υδροφόρους ορίζοντες, επιτρέπει την δίληση του βρόχινου νερού, δίνει στο περιβάλλον τη δυνατότητα ανακύκλωσης και ε, αφομοίωσης των ρήπων σε υδρολογικό επίπεδο. Μιλάμε για μια περιοχή πράσινη, 138.000 τετραγωνικών μέτρων, 14 εκτάρια. Όπως βλέπετε, ακριβώς δίπλα στην περιοχή αυτή, Υπάρχει μια βιομηχανική ζώνη εγκαταλελειμμένη. Ακριβώς στο πλάι, απέναντι. Ε, Ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι διαφορετική η Δήμη, άρα οι αρχέ. Εμεί έχουμε έρθει εδώ διότι η κοντοφθαλμιοπροσέγγιση προσέγγιση των αρχών μα δεν έχουν ανακηρύξει την περιοχή αυτή ω προστατευόμενη. Εδώ όμω νομίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να δει το πράγμα με μια πλέον ε, ε, με μια περισσότερο διορατική προσέγγιση και να πει εάν θέλουμε να επιδιώξουμε τους στόχους ε, καταπολέμησης της ρήπανσης, καταπολέμησης της χρήσης του τσιμέντου παντού, να μια επιφάνεια που πρέπει να προστατευτεί. Πάει ακριβώς στη σωστή κατεύθυνση. Να τι έλεγε η Επιτροπή το 2011. Αυτά έλεγε. Και εμεί το ίδιο λέμε. Επαναλαμβάνουμε τα λόγια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εσεί τα είπατε πριν 8 χρόνια. Αυτό ζητάμε τώρα. Όχι τίποτα άλλο. Αυτό είναι μια διαφάνεια που αποδεικνύει το ποσοστό χρήσης του εδάφους για αστικούς σκοπούς. Πάντοτε προς την κατεύθυνση να μειώσουμε για να μην μπορούμε να μηδενίσουμε την χρήση του εδάφους. Έχουμε 60% χρήση του εδάφους για αστικούς σκοπούς στην στέγη και κατοικία στην περιοχή μας. Αλλά η ίδια σύγκριση ισχύει εδώ, όπως αυτή που κάναμε πριν με την ρήπανση. Αν δούμε τα προγράμματα, τα σχέδια της τοπικής κυβέρνησης που περιγράφουν την πολεοδομική ανάπτυξη που προβλέπεται για τους Δήμους και τις κοινότητέ μας, λένε ότι εντό των έργων αυτών προβλέπεται αύξηση της χρήσης του εδάφους κατά 61,2%. Ε, ε 61,5%. Η ερώτηση λοιπόν είναι, πάμε στην κατεύθυνση που ανέφερε και ανακοίνωνε η ίδια Επιτροπή το 2011 ή μήπως έχουμε πάει σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Εδώ υπάρχει και ένα βίντεο, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείξετε. Να ένα σύντομο βίντεο το οποίο γυρίσαμε για να καταλάβετε γιατί έδαφος μιλάμε. Λέμε 14 εκτάρια. Δείτε εκεί στο βάθος αυτή είναι η βιομηχανική ζώνη εγκαταλελειμμένη. Μιλάμε για περίπου 100 μέτρα απόσταση μεταξύ των δύο περιοχών. Αυτή είναι η έκκλησή μας και είναι ξεκάθαρη. Σταματήστε αυτό το έργο. Τίποτε άλλο. Δεν έχουμε καμία άλλη απέτηση πάει ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η περιφέρεια της Λομαρδίας ανακοινώνει από χρόνια. Μείωση της χρήσης ε, του εδάφους για σκοπούς ε, αστικούς και μείωση της ρήπανσης, της ατμοσφαιρικής κυρίας, κυρίως που έχει να κάνει πάνω απ' όλα με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Ευχαριστώ και με συγχωρείτε που καθυστέρησα. Ευχαριστώ και για πέντε λεπτά ο λόγος στον κύριο Μαουρίτσιο Τσινέζη. Ευχαριστώ. Buongiorno. Buongiorno. Καλημέρα. Εμείς ε, στο Τσινιζέλο Μπάλσαμο είμαστε σε μια κατάσταση όπου ξεκινούν οι εργασίες για ένα εμπορικό κέντρο το οποίο είχε κλείσει στην αρχή ε, λόγω έλλειψης ε, πελατών είδε μια ανάπτυξη όπως είπαν και οι συνάδελφοι και έχουμε εδώ πέρα δύο πολύ σημαντικέ ε, πτυχέ. Εγώ θα προσπαθήσω να ρίξω βάρο ε, στο θέμα των μεταφορών. Το εμπορικό αυτό κέντρο περικλείεται από τέσσερις πολύ σημαντικές οδούς. Ε, τον Α52, τον Α4, τον SS36 και τη Βία Βαλτελίνα. και βεβαίω η κατάσταση των μεταφορών είναι καθημερινά τραγική. Μόνο στο δρόμο 36 που συνδέει το Μιλάνο με το ΕΚΟ έχουμε κάθε μέρα 360.000 ε, διελεύσεις οχημάτων το χρόνο. Βλέπετε τι γίνεται τις ώρες εχμής. Το βλέπετε εδώ πέρα. Συγγνώμη. Να το. Βλέπετε ξεκάθαρα ότι στους τέσσερις αυτούς δρόμους ε, έχουμε διέλευση πάνω από 3.000 οχήματα την ε, ημέρα και η κατάσταση είναι ήδη ε, πολύ κακή. Αυτή είναι η κατάσταση εδώ και η τοποθεσία των εμπορικών κέντρων που υπάρχουν στην ε, περιοχή στο Τσινιζέλο Βάλσαμο το κίτρινο και το Σέστο Τζαντζοβάνι επίσης που έχει δει τρομερή ανάπτυξη 200.000 ε, τετραγωνικών μέτρων ε, έχουμε ένα κέντρο υγείας πανεπιστημιακό νοσοκομείο δηλαδή τεράστιο στην περιοχή αυτή έχουν προβλεφθεί να περνάνε ένα εκατομμύριο άτομα την ημέρα. Γιατί ε, θα πρέπει να φτάνουν στην, ε, στο κέντρο του Μιλάνου ε, και έχουμε βεβαίω την ε, γραμμή του μετρό η οποία έχει καθυστερήσει πέντε χρόνια. Και αν ε, έρθουν και αυτοί οι άνθρωποι προς την γραμμή του μετρό δεν θα βρουν να παρκάρουν. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα την ευρύτερη περιοχή όπου διακρίνεται ξεκάθαρα ότι ο δρόμος 36 που μας ε, συνδέει με τον SP5 θα μπορούσε να βοηθηθεί όσο υπάρχουν έργα στους ε, άλλους δρόμους αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν καταφέρνουν να ξεκινήσουν τα έργα στους άλλους ε, δρόμους. Το τσινιζέλο μπάλσαμο βλέπει, έχουμε εδώ πέρα 10 χρόνια καθυστέρησης, παραδείγματος χάρη ο δρόμος ο 35 θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κάλλιστα για να μην περνάνε οι άνθρωποι μέσα από το τσινιζέλο μπάλσαμο. Αλλά έχουμε τον 36, έχουμε κάνει και κάποιες σχετικές ερωτήσεις. Θα έπρεπε να έχει υλοποιήσει μια υπόγεια διάβαση, αλλά αυτό δεν γίνεται καθόλου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν Ε, έχουμε μία λεωφόρο που οδηγεί στους άλλους δρόμους. Εν ολίγης. Τα, τα αυτοκίνητα θα μας θάψουν. Σε μία προσωμείωση που έχει κάνει το Πολυτεχνείο του Μιλάνου βλέπουμε ότι από το 7 στο 9, ως το 9% των αυτοκινήτων θα παραμείνουν μπλοκαρισμένα και δεν θα καταφέρουν ποτέ να φτάσουν στον ε, προορισμό τους. Επιπλέον, έχουμε κατά μέσο όρο 6.000 άτομα την ε, ώρα, τα οποία φτάνουν με το μετρό μη ένα και προβλέπεται και άλλο ένα το οποίο θα φτιαχτεί λέει το 2030 την πρώτη γραμμή του μετρό. Οπότε ζητάμε εδώ πέρα τέσσερα απλά πράγματα. Το πρώτον, η ευρωπαϊκή κοινότητα να δει τα τέσσερα ερωτήματα που έχουμε κάνει το 2013, τις τέσσερις προσφυγές για τις οποίες ακόμα περιμένουμε κάποια απάντηση. Λοιπόν, ε, το θέμα είναι κρίσιμο όσον αφορά το σταμάτημα των ε, εργασιών γιατί ε, συνεχίζουν και τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα γιατί προβλέπουν 157 φορτηγά τριαξονικά τα οποία θα μετακινούν τα υλικά. Και εντωμεταξύ ο Υπουργός Μεταφορών της Ιταλίας πρέπει να βρει ένα σχέδιο Β για να αποφευχθεί το απόλυτο μπλοκάρισμα της ε, κίνησης. Επιπλέον για την υγεία πρέπει να γίνει επιτέλους μια επιδημιολογική μελέτη στην ε, ζώνη αυτή. Πρέπει να ξέρουμε, πρέπει να καταλάβουμε ποιοι πεθαίνουν, πόσοι πεθαίνουν, γιατί πεθαίνουν, εάν θέλουμε πραγματικά να καταλήξουμε σε μια λύση. τα εμπορικά κέντρα είναι μια πραγματικότητα και υποκαθιστούν τα εργοστάσια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και χρήσιμα. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και να δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για να μας εκθέσει την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπατε, η κατάσταση στην κοιλάδα του Πάδου είναι κάτι που γνωρίζουμε. Έχουμε δύο επιπαραβάσεις διαδικασίες εξέλιξη. Η μία εξετάζεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η Ιταλία έχει ήδη παρουσιάσει τις ε, δικές, τα δικά της στοιχεία ως υπεράσπιση από το 2010 και μετά και όπως έδειξε και ο χάρτης της διαφάνειας, η κοιλάδα του Πάδου είναι από τις πιο μολυμένες περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, από πρώιμου, πρόωρους θανάτους, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την ατμοσφαιρική ρήπανση. Έχει ένα θλιβερό ρεκόρ εδώ η Ιταλία του μεγαλύτερου αριθμού θανάτων που έχουν να κάνουν με τη ρήπανση από μικροσωματίδια. 60.000 θάνατοι ετησίως. Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι 5.000 ο μέσος όρος. Όλα αυτά ε, έχουν άμεση σχέση με την ε, σφαγή που προκαλεί, μπορεί να το πει κανεί, ε, τι μαζικέ απώλειε προκαλεί η ατμοσφαιρική ρήπανση. Είναι πάρα πολλέ περιπτώσει όπου θα πρέπει να ασχοληθώ με το θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το καθένα από αυτά τα έργα που συμπεριλαμβάνει η αναφορά αυτή παρουσιάζει τι δικέ του δυσκολίε. Πρέπει να δούμε ποιο είναι το ευρύτερο πλαίσιο. Μιλάμε για περιοχέ ιδιαίτερα χτισμένε με ανυπόφορα επίπεδα ατμοσφαιρική ύπαρξη. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σύντομα θα αποφανθεί και το δικαστήριο θα αποφασίσει αν έχουμε δίκιο να πούμε ότι το, τα σχέδια των ε, περιφερειών της Λομπαρδίας, του Βένετο ή του Πιεμόντα και άλλων ε, είναι ασύμβατα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Αν όμως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβεβαιώσει ότι το πρόγραμμα για την ποιότητα της του ατμοσφαιρικού αέρα της Λομπαρδίας δεν είναι κατάλληλο, τότε τα έργα αυτά θα πρέπει να τα δούμε από άλλη σκοπιά και να διορθωθούν. Διότι από το 2010 που έχει ανακυρωχθεί η ζώνη αυτή ε, για την... Ε, ε, υγεία λόγω της ατμοσφαιρικής ρήπανσης δεν είναι η μόνη που δεν έχει κάνει τίποτα. Η κοιλάδα του Πάδου έχει πάρα πολύ δύσκολε συνθήκε και χειροτερεύουν το 2010. Φανταστείτε ότι με τι ιδιαιτερότητές τη αυτό που συμβαίνει είναι λες και είμαστε καπνιστές και βρισκόμαστε σε ένα κλειστό δωμάτιο χωρί να ανοίγουμε ποτέ τα παράθυρα και καπνίζουμε πολύ μαζί. Ενώ σε άλλε περιοχέ ε, ο αέρας μπορεί κάπως ε, κάπως καταφέρνουν να ε, καθαρίσουν τον αέρα τους ε, σε άλλες γεωγραφικές περιοχές. Θα μπορούσε να είναι αδιάφορο το τι συμβαίνει συνολικά. Αλλά στην κοιλάδα του Πάδου βρισκόμαστε σε ένα δωμάτιο που καπνίζουμε χωρίς παράθυρα. Αυτό γίνεται διαρκώς κάτι που προκαλεί ε, σοβαρά προβλήματα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχουμε εργαλεία για την χρήση του εδάφους που σωστά αναφέρθηκε δικαίως ότι χρειάζεται μια πώληση, μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2011 που προέβλεπε ότι θα υιοθετηθούν υποχρεωτικές δεσμευτικές πράξεις ε, για την ε, ε, χρήση του εδάφους και την ε, γυτνίαση με τον άλλο βιομηχανικό χώρο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα δυστυχώς. Θα έπρεπε να υπάρχει μια πράξη, κάτι δεσμευτικό, μια οδηγία, μια απόφαση. Για αυτό το θέμα λοιπόν σημειώνω παραβίαση της οδηγίας που αναφέρθηκε στην περίπτωση του Αρέζε συγκεκριμένα. Στην περίπτωση του Αρέζε μαθαίνουμε σήμερα ότι απορρίφθηκε, μάλλον έκλεισε το γραφείο που συγκέντρωνε στοιχεία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Αυτό ε, παραβιάζει το άρθρο 5 της οδηγίας, όπου ορίζεται και μπορώ να αναφέρω και να παραθέσω ε, το εδάφιο, μισό λεφτάκι, γιατί έψαχνα ενώ σας άκουγα. τα σημεία δειγματοληψία που δείχνουν ότι υπάρχει υπέρβαση των μέσων αξιών των τελευταίων ετών πρέπει να καταγράφονται. Δεν μπορεί λοιπόν να κλείνει ένα γραφείο ε, Εκεί που φαινόταν ότι υπήρχαν υπερβάσει αμέσω την προηγούμενη χρονιά, όταν συνέλεγε στοιχεία, η περίπτωση του Αρέζα λοιπόν αποτελεί πρόδειλα ε, περίπτωση πιθανή παραβίαση και το καταγράφουμε. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα και εκεί κάτι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Για τα υπόλοιπα στοιχεία τη αναφορά πρέπει να λάβουμε υπόψη το γενικότερο πλαίσιο. Η κοιλάδα του Πάδο έχει σοβαρότατα προβλήματα ρήπανση από το 2010 με διοξίδιο του αζότου, πάρα πολύ ανησυχητικά επίπεδα και τιμέ. Ε, είναι πολύ ανησυχητικό το τι γίνεται και με τι δύο προηγούμενε παραβιάσει που ανέφερα. Οπότε ε, θα συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε διότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για τα επιμέρους εμπορικά κέντρα, αλλά μπορούμε να κάνουμε κάτι συνολικά, ε, ίσως για τη συνολική συμμόρφωση. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ, πολύ ξεκάθαρη τοποθέτησή σας. Και τώρα οι συνάδελφοι, κυρία Εύη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους αναφέροντες οι οποίοι μας παρουσίασαν μια κατάσταση που πραγματικά μας κάνει να ανησυχούμε ιδιαίτερα δραματικά για την περιοχή του Μιλάνου, ιδίως στα βόρεια της πόλης. Ε, υπάρχει πολεδομικό σχεδιασμό στην περιοχή που δεν κάνει άλλο παρά να οδηγεί την, ε, σε αύξηση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης και σε κακή χρήση του εδάφους και περισσότερο χτίσιμο της περιοχής, ε, τη του τσιμέντου. Οι ανησυχίε που εξέφρασαν λοιπόν οι αναφέροντε, αυτά που μα είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ η ίδια, ε, είναι πράγματα που τα καταγγέλλω εδώ και χρόνια. Το θέμα τη ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, τη ατμόσφαιρα στην Ιταλία, στην Λομβαρδία, γενικώ είναι πλέον δομικό. Ε, όμως, ε, επειδή έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις επιτόπου και κάποιος προγραμματισμός εδώ τοπική, περιφερειακής κυβέρνησης ε, για το θέμα αυτό, μόνο χειρότερα πάνε τα πράγματα. Τα δεδομένα που μας παρουσίασαν οι αναφέροντες και η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα επιβεβαίωσε με τη σειρά τη, είναι δεδομένα ε, που προκύπτουν από τη δουλειά των εκθέσεων, των μελετών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Είναι δραματικά τα στοιχεία. Η Ιταλία έχει πραγματικά ένα πολύ θλιβερό ρεκόρ ε, πρόωρων θανάτων λόγω της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το σημείο. Θέλω να υπογραμμίσω, όπως είπαν και οι αναφέροντες, ότι υπάρχει επιδείνωση, περαιτέρω ε, υποβάθμιση της κατάστασης και αύξηση των πρόωρων θανάτων ε, λόγω ατμοσφαιρικής ρήπανσης και των καρδιαγγειακών παθήσεων, που ήδη έχουν καταγραφεί και εξαιτία τη εκτέλεση των έργων αυτών στην περιοχή. Καταγράφω με ιδιαίτερη ανησυχία και εγώ ίδια το γεγονό ότι έκλεισε εκείνο το γραφείο ε, σε μια από αυτέ τι κοινότητε, το Αρέζε. Είναι σαφή παραβίαση, κατάφορη παραβίαση των όσων ε, ορίζει οδηγία. Οπότε θα πρέπει να ανοίξουμε και να περάσουμε στις νόμιμες οδούς για να ξεκινήσει η διαδικασία που παραβάσει. Αλλά είναι ένα πρόσθετο στοιχείο πολύ, πολύ σοβαρό. Διότι αν σήμερα όποιος έχει την αρμοδιότητα να προστατεύει την υγεία των πολιτών και υποχρεούται να καταγράφει στοιχεία, να παρακολουθεί το τι συμβαίνει με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και αυτό γίνεται κάποιε φορέ το ή άλλω με αλλίωση των στοιχείων, γιατί είναι ιδιώτε αυτοί που αναλαμβάνουν την καταγραφή του ή σε κάποιε περιοχέ τα γραφεία ε, πάνε σε ε, περιοχές της υπαίθρου, οπότε πού να καταγράψουν σωστά την ποιότητα ε, του ατμοσφαιρικού αέρα. Βρισκόμαστε εν μέσω του παραλόγου κάτι το παράδοξο, όπω το γεγονό ότι έκλεισε αυτό το γραφείο. Είναι ένα γεγονό που είναι ε, μεγάλη σοβαρότητα, είναι ανήκουστο και δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε. Γι' αυτό λοιπόν να κλείσω λέγοντα ότι πρόσφατα επέβαλα και προφορική ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κατά πόσον το πρόγραμμα για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην περιοχή τη Λομβαρδία ε, έχει προχωρήσει και αν προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα τη ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Εδώ είναι γεγονό ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο Προσπαθούμε να κάνουμε περισσότερα. Την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλεια συζητήσαμε την σημαντικότατη πρωτοβουλία του Ευρωκοινοβουλίου που υποστήριξε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρχουν πράσινε περιοχέ για όλου. Αυτή είναι η κατεύθυνση που θέλουμε να ακολουθήσουμε και είναι απαραίτητο να αλλάξουν τελείω ε, το πώ λειτουργούν όλοι οι κλάδοι που προκαλούν ρήπανση. αυτό των οδικών μεταφορών, που μας ανησυχεί πάνω από όλα αυτή τη στιγμή, ιδίω κοντά σε αστικέ περιοχέ. Γι' αυτό λοιπόν τέτοιου είδου έργα τεράστιων διαστάσεων είναι ιδιαίτερα επιζήμια για τι περιοχέ που κατοικούνται κιόλα. Εδώ υπάρχουν τεράστιε ευθύνε σε επίπεδο τη περιφέρεια τη Λομβαρδία που είναι κοντόφθαλμη. Δεν σταμάτησε, δεν ανέκοψε την πορεία τέτοιων έργων και την εκτέλεσή του. σα ίσα τα πρημοδοτεί και εδώ να κάνω και μια αναφορά στη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οργανώσαμε και μια ακρόαση με τη συμμετοχή της Επιτρόπου Μπιανκόφσκα ε, και η έκβαση, τέλος πάντων η παρακολούθηση του τι έγινε μετά τον Dieselgate. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι βιώσαμε ένα σκάνδαλο που ακόμη και σήμερα μας καίει. Ε, είναι ανοιχτή το θέμα. Είναι εκατομμύρια επί εκατομμυρίων τα οχήματα που κυκλοφορούν στου αυτοκινητοδρόμου και του δρόμου τη Ευρώπη και μολύνουν πολύ περισσότερο, ε, ρηπαίνουν πολύ περισσότερο από ό,τι είχε αναγγελθεί, από ό,τι προβλεπόταν. Και το πρόβλημα αυτό ακόμα δεν έχει επιληθεί. Δεν έχουν γίνει αρκετά. Ούτε έχουν βρεθεί τα καταλληλότερα και δραστικότερα μέτρα. Έχουμε δύο ε, κολάφους ε, που είναι πραγματικά ηχηρίω προ προς την υποτιθέμενη δράση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής για να επιλύσει το θέμα αυτό, αποφάσισε του Ευρωπαϊκού δικαστήριο που δείχνει ότι ο διπλασμό των ορίων για το διοξείδιο του αζότου είναι προφανές ότι απλώς φάνηκε να λύνει το πρόβλημα, αλλά από την άλλη υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου λόγω των προσφυγών κάποιων κοινοτήτων και δήμων, αρχών τοπική αυτοδιοίκηση, μεταξύ των οποίων η πόλη τη Μαδρίτη, του Παρισιού και του καταξή, που ζήτησαν από το δικαστήριο βοήθεια. Ζήτησαν βοήθεια ακριβώ για να προβλεφθεί ένα παράγοντα συμβατότητα, συμμόρφωση που να περιγράφει επιτρέπει στους παραγωγούς να μην βγάζουν πάλι στα οχήματα, να μην βγάζουν στους δρόμους οχήματα που ρηπαίνουν ακόμη περισσότερο από ό,τι προβλέπουν τα όρια των ευρωπαϊκών οδηγιών που πρέπει να εφαρμόζονται. Κλείνω λοιπόν εδώ. Οι ευθύνε είναι πολλών είναι κοινέ, αλλά αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι η περιφέρεια τη Λομπαρδία πρέπει να κάνει περισσότερο και να σταματάει τα έργα αυτού του είδου. Αυτέ οι αναφορέ να συνεχίσουν να εξετάζονται, αυτή είναι η δική μου σύσταση, βάσει των παραβιάσεων που ούτω ή άλλω βλέπουμε ότι εξετάζονται, μα το είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και πρέπει οι αναφορέ αυτέ να απευθυνθούν και στην ίδια την περιφέρεια, την περιφέρεια της Λομπαρδίας και θα πρέπει να αποσταλούν και στο Δήμο, στις δημοτικές αρχές και στις κοινότητες ε, ή όσους έχουν εγκρίνει την οικοδόμηση των ε, εμπορικών αυτών κέντρων στο Αρέζε, το Τσινιζέλο Μπάσαλμο και το Μπολάτε. Ε, θα πρέπει επίσης να απευθυνθούμε και στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Υγείας διότι ξέρω ότι δίνουν μάχη και σε αυτό το μέτωπο, ιδίως με το Cleaner ε, Dialogues που ε, ξεκίνησαν στο επίπεδο των διάφορων δήμων και περιοχών γύρω από την κοιλάδα του Πάδου, αλλά πρέπει να τους ανα... Ε, ενθαρρύνουμε να κάνουν περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν τους αναφέροντες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα στοιχεία που μας έδωσε. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποιος άλλος? Όχι. Λοιπόν, νομίζω ότι η κατάσταση είναι σαφής. Ε, κρατάμε νυχτέ και τις τρεις αναφορές. Στηρίζουμε τις δραστηριότητες της Κομισιόν. Ε, καλό είναι να περιμένουμε τα αποτελέσματα της, ε, των διαδικασιών εκ παραβάση και κυρία Αέβη, κατόπιν του ετοιματός σας νομίζω θα στείλουμε κάποιες επιστολές στις Ιταλικές ε, Περιφερειακές Αρχές και στο Υπουργείο Υγείας στην Ιταλία. Εντάξει, το δέχεστε. Ωραία, σε ευχαριστώ. Ωραία, θα συνεχίσουμε οπωσδήποτε τον διάλογο μας ε, και στο μέλλον ε, όταν θα έχουμε νεότερες πληροφορίες από την Κομισιόν. και από τις Ιταλικές Αρχές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να δώσετε πάλι το λόγο στους ε, αναφέροντες για ένα σύντομο σχόλιο. Αν θέλουν βεβαίως. Σύντομα. Θα ήθελα να πω κάτι σύντομα. Ακούσα τον κύριο της Κομισιόν που χρησιμοποίησε μια περίεργη έκφραση. Νομίζω δεν θέλαμε να το χρησιμοποιήσουμε γιατί είναι κάπως υπερβολικό, αλλά δεδομένου των αριθμών που γνωρίζουμε, πραγματικά πρόκειται περί σφαγής. Το θέμα το οποίο Ε, Μα ανησυχεί εδώ πέρα είναι πώς τελειώνει μια διαδικασία επί παραβάση ή μάλλον όσο καιρό θα διαρκεί θα έχουμε 5.000 πρόωρους θανάτους το μήνα. Κάθε μήνα που περνάει χάνονται άνθρωποι. Το πρώτο θέμα λοιπόν, η πρώτη αμφιβολία μας προωρους τους ακριβώς ότι από όσο ξέρω η πρώτη διαδικασία ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια. Όχι, όχι. Παρ' αυτά ε, θέλω να καταλάβω το χρονικό πλαίσιο γιατί αν μιλάμε μόνο για πρόστιμα χωρίς ε, να υπάρχει κάποια δυνατότητα παρέμβασης επίσης για την ε, μέτρηση ακούσαμε ότι λείπουν μια σειρά σταθμών κέντρησης και το μόνο κέντρο το οποίο υπάρχει στην περιοχή μας ε, είναι σε μια γειτονική περιοχή. Αλλά θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει και μια παρέμβαση για να βελτιωθεί η κατάσταση. Αλλιώς θα συνεχίσουμε απλά να μετράμε ε, τους θανάτους. Ε, δεν είναι λύση αυτό το πράγμα. Ανησυχητικό είναι επίσης ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρέμβει σε μια τέτοια περίπτωση. Γιατί πάντα έτσι θα γίνεται. Οι περιφέρειες κοιτάνε πρώτα την οικονομική πτυχή και μετά την ε, πτυχή της υγείας. Ε, είναι όμως μια ευρωπαϊκή, είναι ευρωπαϊκό δικαίωμα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις μικρές, ε, γιατί βλέπετε εδώ πέρα και αυτές μικρές είναι, αλλά μία-μία μαζί καταλήγουν σε μια κατάσταση δραματική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για το χρονοδιάγραμμα. Θα απαντήσω τελικά. Ε, Έχετε δίκιο όταν ε, λέτε ότι χρειάζονται μεγαλύτερη χρόνοι για τόσο περίπλοκε υποθέσει. Περιμένουμε απόφαση όμω εντό τη ε, χρονιά. Διότι έχει λήξει η προθεσμία η Ιταλία υποβάλει τα στοιχεία της υπερασπισή της. Θα πάμε σε πραγματική διαδικασία στο Λουξεμβούργο σύντομα ε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η Ιταλία έχει ήδη καταδικαστεί το 2010 για τα θέματα αυτά. Επ' αυτού. Ε, πέρα της κουβέντας ε, για τις πινακί... για, για τα πρόστιμα και τις του πίνακε που του ε, ξανακοίταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χθε για να προσαρμόσει τα ποσά, ξαναείδαμε και διορθώσαμε το τι θα γίνει με το θέμα. Ε, αλλά αυτό που μπορούσε να το έχει κάνει η Περιφερεια τη Λομβαρδία εδώ και πολλά χρόνια γιατί γνώριζε πάρα πολύ καλά τη σοβαρότητα τη κατάσταση. Κατά την άποψή μα, ε, όσα προβλέπονται ω τώρα ω ε, προγράμματα είναι τελείω παράδεκτα, αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αν θα προχωρήσει εγκαίρω για να εκδοθεί η κατάλληλη απόφαση. Σα ευχαριστώ και φυσικά θα συνεχίσουμε στο μέλλον το διάλογο μας, στο μέτρο που λαμβάνουμε νέες πληροφορίες. Ευχαριστώ και περάμε στο τελευταίο σημείο, αν δεν κάνω λάθος, της ε, ημερήσιας διάταξής μας. είναι ε, τα επικίνδυνα χρηματοπιστωτικά μέσα στην Ισπανία, στις Ισπανικές τράπεζες. Έχουμε πάνω από 20 αναφορές ε, και έχουμε παρόντες εδώ δύο υποβάλλοντες αναφορά, την κυρία Στέβεση Ροντρίγκες και το Χεσούς Δομινίκες. Ντομίνγκες και Ροντρίγκες, συγγνώμη. Είναι σωστές οι πληροφορίες μου. Κύριε Ροντρίγκε, Χωσέ Μανουέλα Στέβε Ροντρίγκε, έχετε πέντε λεπτά για να μα παρουσιάσετε την αναφορά σα. Καλημέρα σα καταρχήν. Πριν από 7 χρόνια, το 2012, υποβάλαμε μία αναφορά κάνοντας μία καταγγελία για δόλιες τραπεζικές πρακτικές. Και μάλιστα τεκμηριώσαμε την αναφορά μας ε, με επαρκή έγγραφα που αποδεικνύουν πόσο απατηλό και δόλιο ήταν το σύστημα, όχι μόνο στη συγκεκριμένη τράπεζα, αλλά σε 52 από τις 56 τράπεζες της Ισπανίας. Ήταν καταχρηστικές και ε, χροκερδείς αυτές οι πρακτικές. Η απάντηση που μου δώσετε ήταν μια ανακοίνωση προς τα μέλη, στην οποία αναφέρονται οι περιλήψεις των 22 αναφορών. Στη σελίδα 8 αναφέρεστε στο άρθρο 216 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λέτε ότι οι ιδεοντολογικοί κανόνες για την καταλληλότητα, τη, την ειδωλιότητα, τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη κατοχυρώνται στην οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, τη MIFID. Και θα πρέπει να δίνεται το καλύτερο προϊόν στον κάθε ε, πελάτη ανάλογα με τις προσωπικές του συνθήκες και τα συμφέροντά του. Δηλαδή, αυτά που αναφέρεται παραπέμπουν στη MIFID. Έχουμε και το 2004-39, τον 1287 ε, κανονισμό και εκεί αναφέρονταν η προστασία του καταναλωτή του πελάτη. Οι συγκεκριμένε διατάξει ενισχύονται με τι νέε κατευθυντήριε γραμμέ για τα εφαρμοστικά μέτρα. Αυτό που λέμε μεταφορά των οδηγιών. Στην ε, οδηγία 8 της ανακοίνωσης ε, αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ε, επιβλέπει τη σωστή μεταφορά και σωστή εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να εξετάσει περιπτωσιολογικά κάποιε καταστάσει. Αλλά όταν 52 από τι 56 τράπεζε ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τη ε, χώρα ε, παραβιάζουν την νομοθεσία και όταν περίπου ένα εκατομμύριο Ισπανοί πολίτε ε, πλήττονται από αυτή την ελλειπή μεταφορά τη οδηγία, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια στιγμή να παρέμβει. Παρ' όλα αυτά δεν το κάνει. Μάλιστα, ε, αναφέρονται οι ενισχυμένες διατάξεις για την κατάσταση των καταναλωτών, εμ, αναφέροντας κάποια μέσα που δεν καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύης Καταθέσεων και ότι δεν θα πρέπει να δίνονται αυτά τα χρήματα στους ε, εμ, ιδιώτες επενδυτές. Αλλά μπερδεύεται τον επενδυτή με αυτόν που κάνει αποταμίευση. Άλλο κάποιο που έχει οικονομίε και τι αποταμιεύει και άλλο επενδυτή. Δεν θα πρέπει να εξομοιώνεται τι δύο έννοιε. Πρόκειται για ιδιώτε που προσπαθούν, ε, νομίζαν ότι αποταμίευαν τα χρήματά του και στην ουσία ε, εξομοιώνονταν με επενδυτέ. Εμένα με εξαπάτησαν λέγοντας ότι οι οικονομίες ε, ολόκληρης της ζωής μου ήταν ουσιαστικά μια κατάθεση και μέσα σε 24 ώρες θα μπορούσα να κάνω ανάληψη. Και δεν εξαπάτησαν μόνο εμένα, αλλά και ένα εκατομμύριο συμπολίτε μου. Γι' αυτό και θα πρέπει να ζητήσετε, να απαιτήσετε από την κυβέρνηση της Ισπανίας ε, να πληρώσει αυτό το χρέος της προς τους ε, πολίτες που έχουν ε, πληγεί. Μάλιστα, η η Τράπεζα Χιμένες έδωσε 2009 στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα κείμενο που λέει ότι όλοι είναι επενδυτές με εξαίρεση μία μικρή ομάδα που έκαναν ε, ε, οικονομίες και έκαναν την αποταμίευσή τους. Ουσιαστικά δηλαδή μας λέει όλους οι επενδυτές. Ελάχιστοι είναι αυτοί που χαρακτηρίζονται ως αποταμιευτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι θα πρέπει να αναλάβουμε ένα γραμμάτιο και να γίνει μια κατανομή του χρέους μεταξύ όλων των ε, Είναι απαράδεκτο να έχει περάσει μία επταετία και ακόμη να κρεμεί η διαθέτηση αυτού του ζητήματος. Πάνω από 200.000 ε, αιτήσει έχουν υποβληθεί για διατησία και 100.000 τέτοιε αιτήσει έχουν γίνει δεκτές και έχουν διεκπεραιωθεί όλες οι αποφάσεις της διατησία δικαίωσαν τους ε, προσφεύγοντε Στι περισσότερε καταγγελίε δικαιώθηκαν οι προσφεύγοντες και εσεί μα λέτε ότι το θέμα της σωστής μεταφοράς ανήκει στην ισπανική δικαιοσύνη. Εδώ δεν μιλούμε για μία-δύο περιπτώσεις. Εδώ μιλούμε για ένα εκατομμύριο πολίτες που έχουν πληγεί. Δεν θα πρέπει να επαναληφθεί μια τέτοια κατάσταση, θα πρέπει να διορθωθεί. Αυτό που συνέβη με τις υποθήκες σε λίγο θα γίνει με τις πρόορες συντάξεις, με τους συνταξιούχους, με τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Αν πραγματικά θέλουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες, τους εργαζόμενους, θα πρέπει να αλλάξουμε την νομοθεσία. Δεν μπορούμε να ερχόμαστε εδώ ε, να κάνουμε μια καταγγελία και μετά από μια πταετία να βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο, να μην έχει αλλάξει τίποτα. Και μάλιστα έγινε συγχώνευση δύο τραπεζών ταμιευτήριων ε, λόγω της τεχνικής πτώχευσης στην οποία ε, βρισκόταν. Και μάλιστα χρησιμοποίησε πολύ επιδέξια έναν εξωτερικό έλεγχο, που ήταν ουσιαστικά μια έκθεση και μάλιστα καταβλήθηκε ένα εκατομμύριο ευρώ για την εκπόνηση αυτής της μελέτης και ο κύριος Χουέγος και η κυρία Μάρτα Φουέρας ισχυρίζονται ότι μέσα σε μία χώρα θα δίνουν και κέρδη αυτές οι τράπεζες μετά τη συγχώνευσή τους. Έτσι όμως πτώχευσαν δύο τράπεζες της Γαλλικίας. Το 2011 ε, αναφέρεται σε μία έκθεση όπου πολιτικά κόμματα της Γαλλικίας, ε, οι τράπεζες της Γαλλικίας χρωστάνε 500 εκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες αυτές. Και αυτά τα 515 συγκεκριμένα εκατομμύρια ευρώ τελικά επιστράφηκαν ε, στα χρηματοπιστωτικά αυτά ιδρύματα ή είναι η βάση ώστε τα τα πολιτικά κόμματα και οι τοπικοί φορείς ε, κάνουν την πάπια και αφήνουν 75.000 οικογένειες χαλικίες να χάνουν τις οικονομίες τους ολόκληρες ή ένα τμήμα τους. Δεν αρκεί προσφυγή στα δικαστήρια. Θέλουμε μια απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχήν, να γίνει μια διάγνωση της κατάστασης, μια διαπίστωση της κατάστασης και μετά να βρεθούν λύσεις για να αποφευχθεί επανάληψη μια τέτοια κατάσταση και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ο... κυρία για πέντε λεπτά. Ο κύριος Ντομίγκες, συγγνώμη, για πέντε λεπτά. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας που κράτησε ανοιχτή τη συγκεκριμένη αναφορά. Έχουμε και μία σύντομη έκθεση, ένα δελτίο τύπου και διάφορα άλλα έγγραφα, ώστε να εξαλείψουμε αυτές τις ε, καταχρηστικές πρακτικές πολλών ισπανικών τραπεζών. Όταν καταθέσαμε την αναφορά μας, είχαμε επίγνωση ότι η πρωταρχική ευθύνη ήταν των τραπεζών. Αλλά τέτοιε καταχρηστικές πρακτικές δεν θα ήταν ε, δυνατόν να υλοποιηθούν χωρίς τη συγκατάβαση ή την ανοχή των ε, αρμόδιων ε, αρχών. Ουσιαστικά όμως έτσι χάθηκαν 42 δισεκατομμύρια ευρώ από οικονομίες λόγω απατών, χωρίς συγκατάθεση και χωρίς κατάλληλη ενημέρωση των, των καταθετών και μάλιστα με παράβαση, παραβίαση της ενωσιακής νομοθεσίας. Στην αρχή οι αρμόδιες αρχές επέτρεψαν την δημιουργία φορολογικών παραδείσων και μετά νομοποίησαν την κεφαλαιοποίηση των εταιριών αυτών με περίπλοκα προϊόντα, ουσιαστικά αναγκάζοντας τους καταθέτες να συμμετέχουν στην διάσωση των τραπεζών. 18 δισεκατομμύρια ήταν οι λεπιτεροί και μάλιστα χωρίς καμία νομική βάση από το νοσιακό δίκαιο. Και μάλιστα η ισπανική απάντηση δόθηκε τον Ιούλιο του 2012. Η μόνη λύση που δόθηκε στους κατοίκους Γαλλικίας ήταν ειρηνικές υποδειγματικές διαβουλεύσεις, ε, διαδηλώσεις, γνώμη ε, δείχνοντας όμως μία πυγμή και ζητώντας να δοθεί μία απάντηση από την κυβέρνηση έγιναν διαιτησίες, και, αλλά έχει επιστραφεί μόνο το 5% των οικονομιών. Και ουσιαστικά την κατεύθυνση την έδιναν οι τράπεζες. Επίσης επιβλήθηκε ένας νόμος για, το, για τα επιτόκια με ad hoc μέτρα και το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ισπανίας έκρινε το νόμο αυτό αντισυνταγματικό και κατήργησε μεγάλο τμήμα των διατάξεων. Μάλιστα, τον Φεβρουάριο του 2017 η κυβέρνηση Ραχώη υπέβαλε βέτο σε μία πρόταση της γαλλικιανής κυβέρνησης προκειμένου να επιστραφούν ε, ολόκληρες ε, οι οικονομίες των καταθετών, όπως έγινε στην Ιταλία. Και μάλιστα δυστυχώς ε, οι μεγάλες ισπανικές τράπεζες εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση επιστροφής των καταθέσεων. Εφαρμόστηκε μάλιστα στην ε, ε, Ισπανία η οδηγία 2014 του 59 που κανονικά έπρεπε να τεθεί σε εφαρμογή το 2016. Αν ήταν τόσο απαιτητικό το Eurogroup το έκανε χωρίς νομική βάση γιατί δεν ίσχυε ακόμη αυτή η οδηγία. Επίσης 60 δισεκατομμύρια έχουν χάσει οι Ισπανικές τράπεζες από τη διάσωση και 13 δισεκατομμύρια δόθηκαν από τους κατόχους των ε, των προνομιούχων μετοχών, ενώ ταυτόχρονα οι, οι τράπεζες εξακολουθούν να έχουν δισεκατομμύρια κέρδη. Και παρόλα αυτά καμία τράπεζα δεν καταδικάστηκε για αυτή τη δόλια πρακτική και για αυτή την τεραστίων διαστάσεων απάτη. Ούτε ε, οι νομοθετικές αρχές, ούτε οι αρμόδιοι φορείς ανέλαβαν κάποια ευθύνη. Και όσοι βρίσκονται στι φυλακέ είναι για άλλε δόλειε πρακτικέ και όχι για τι συγκεκριμένε καταχρηστικέ πρακτικέ. Τι είπε λοιπόν η διερευνητική αποστολή ε, του Γαλλικιανού Κοινοβουλίου, που ουσιαστικά είναι έρμεο τη πλειοψηφία του ΕΛΚ στο κοινοβούλιο αυτό. Και σίγουρα μετά την ένεση 9 εκατομμυρίων στην Γαλλικιακή Κάισα πουλήθηκε ε, μόνο για ε, ένα συμβολικό ποσό, ενώ μέχρι το 2017 είχαν προθεσμία. Και μάλιστα σε αυτή την ε, πενταετία από την ιδιωτικοποίηση, τα κέρδη είναι 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Η διαχείριση αυτή ήταν καταστροφική για τον δημόσιο Κορβανά. Και μάλιστα ε, η υποχρεώση των γραμματείων για τους πελάτες ήταν τραγική. Πολλά χρήματα δεν επιστράφηκαν στους κατόχους των προνομίουχων μετοχών και τελικά αυτοί που βρέθηκαν κερδισμένοι είναι οι μέτοχοι των τραπεζών. Ουσιαστικά ιδιωτικοποιήθηκαν τα κέρδη και ε, μοιράστηκαν οι ζημίες. Ταυτόχρονα οι καταχρηστικέ τραπεζικέ πρακτικέ συνεχίστηκαν. Ασύμετρη πληροφόρηση, δόλια πρακτική, οι εξώσει ανήμποροι πολίτες, δεκάδε χιλιάδε άνθρωποι έχασαν τα σπίτια του, 30.000 το χρόνο κατά μέσο όρο οι Ισπανοί υπέστησαν έξωση. Ενώ ε, υπάρχει ένας κανόνας που μιλάει για την έξωση σε περίπτωση μη πληρωμής 3 με 7%. Ενώ στη Γαλλία ε, είναι 20%, στη Γερμανία 10% η αδυναμία πληρωμής. Και μάλιστα έγινε πρόσφατα μία έξωση μίας ε, ηλικιωμένης κυρίας 70 ετών λόγω μίας δόλης καταχρηστικής πρακτικής. Αποτέλεσμα είναι 200.000 ε, πολίτες στη Γαλλικία να έχουν πληγεί από αυτή την ασύμετρη και παραπλανητική πληροφόρηση. Μάλιστα, μια δικαστική απόφαση υποχρέωσε την πολιτες στη Γαλλική να επιστρέψει ε, όλο το ποσό, αλλά σε δευτεροβάθμια απόφαση περιορίστηκε η υποχρέωση αυτή. Ουσιαστικά έχουμε 300.000 αγωγές μέχρι το 2021. Έχουμε swaps σε 2.000 πελάτες και μέχρι το 2018 είχαμε ε, καταδικαστικές αποφάσεις για τα τραπεζικά ιδρύματα. Επίσης, είχαμε 60.000 οικογένειε που είχαν υπογράψει γραμμάτια υποθήκης και παρά τι ε, δικαστικέ αποφάσει που δικαίωσαν τους καταθέτες, καμία κύρωση ή τιμωρία δεν επιβλήθηκε στις τράπεζες. Επίσης, για τα ενυπόθηκα δικαστικά δάνεια που αφορούν ένα εκατομμύριο υποθήκες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι ίσως αυτός ο δείκτης ε, λόγω αδιαφάνειας ε, διαγραφή ενώ τον ίδιο μήνα είχαμε, ε, περιμέναμε την απάντηση του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου. Επίσης είχαμε ή υψηλά επιτόκια ή εφασφαλμένα επιτόκια, ενώ ελάχιστοι πελάτες έχουν επίγνωση αυτών των πρακτικών για να κάνουν τις καταγγελίες τους και να διεκδικήσουν με αγωγές αυτά που κατέθεσαν. Επίσης, ζητούμε από τις δημόσιες αρχές να προασπίσουν τα δικαιώματα των καταναλωτών, των πελατών να υποβληθούν πρόστιμα και ε, κυρώσεις για τις παραπλανητικές αυτές πρακτικές και μάλιστα τα πρόστιμα να είναι υποδειγματικά για να έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα και να γίνει μια μελέτη των ζημιών που προκάλεσαν αυτές οι τραπεζικές απάτες. Γι' αυτό παρακαλούμε την Επιτροπή να κρατήσει ανοιχτή την αναφορά και να ευχηθώ το έργο της Επιτροπής, ε, της Επιτροπής να εξυπηρετήσει το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών ώστε να περιοριστούν οι καταχρηστικές και δόλε πρακτικές. Και όπως είπε ο κύριος Ροδρίγο Ράδο, το πρώην Υπουργό της Οικονομίας που σήμερα βρίσκεται στι φυλακέ για πολλά ζητήματα και τη Μπάνκια μεταξύ άλλων, είπε είναι η αγορά φίλη. Εγώ λέω δεν είναι η αγορά φίλη, είναι κλοπή και λαιλασία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τώρα να ζητήσω από την εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα παρουσιάσει τη θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μιλήσω γερμανικά, γιατί μου είπατε ότι μπορώ να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα, εντάξει. λοιπόν, να ξεκινήσω με ένα σύντομο ερώτημα, γιατί ο πρώτος ε, ε, τον μίλησε για μια έκθεση την οποία δεν έχω λάβει, δεν ξέρω αν μπορείτε να μου την στείλετε μετά την ε, συνεδρίαση. Όπως υπόθηκε ήδη κατά κανόνα εδώ πέρα αναφερόμαστε σε κάποια χρηματοπιστωτικά μέσα στην οδηγία αυτή περί χρηματαγορών. Ξέρετε ότι εγκρίθηκε η οδηγία το 2004 και θέλουμε ακριβώς να ενισχύσουμε την προστασία των καταναλωτών γιατί στην οδηγία αυτή το θέμα είναι παραδείγματο χάρη μια εταιρεία η οποία προσφέρει τέτοιες υπηρεσίες θα πρέπει να δρά πάντα με τρόπο τίμιο, επαγγελματικό και προς το συμφέρον των πελατών της. Όλες οι πληροφορίες και οι ανακοινώσεις περί marketing που απευθύνονται σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες θα πρέπει να είναι απλές, σαφείς και όχι παραπλανητικές. Οπότε, οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι κατανοητές έτσι ώστε ο πελάτης να καταλαβαίνει το είδος και τον κίνδυνο των υπηρεσιών και τον τύπο του χρηματοπιστωτικού μέσου. Αυτά ε, περιέχονταν ήδη στο νομοθέτημα του 2004. Είδαμε όμως πως υπάρχει κάποια ανάγκη βελτίωσης και προτείναμε μια ενίσχυση του, της προστασίας των καταναλωτών και έτσι καταλήξαμε στην οδηγία MIFID 2 όπως λέγεται η οποία εγκρίθηκε το 2014 και είναι σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2018. Οπότε ίσως να μην ισχύει για κάποιες από τις περιπτώσεις που αναφέρατε, αλλά τώρα θα παρατηρήσουμε ε, εάν ε, έχει βελτιωθεί κάτι από τον Ιανουάριο του 2018. Οι νέοι αυτοί κανόνες ε, βεβαίω εναρμονίζονται και με τον έλεγχο καταλληλότητας και Ακριβώς εδώ πέρα πρέπει να υπάρχει μια δήλωση καταλληλότητας η οποία πρέπει να γίνει και μάλιστα πριν ένα τέτοιο ε, μέσο πολιθεί ή αγοραστεί. Θα πρέπει η δήλωση αυτή να εξηγεί γιατί ταιριάζει ακριβώς η σύσταση που γίνεται στον συγκεκριμένο πελάτη και βεβαίω το βάρος δίνεται στην ενημέρωση του πελάτη για το γιατί του προτείνονται τα συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Και βεβαίω θα πρέπει να αντιλαμβάνετε τον τρόπο λειτουργία και τους κινδύνους ε, του κάθε προϊόντος και ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος θα πρέπει να του κάνει τις σχετικές ερωτήσεις. Ε, ποια είναι τα οικονομικά μέσα που έχει στη διάθεσή του, πόσο θέλει να κινδυνεύσει κτλ. Όλα αυτά καθορίζονται επακριβώ. Η δήλωση αυτή η καταλληλότητας λοιπόν πρώτα απ' όλα είναι το γιατί ταιριάζει σε ένα συγκεκριμένο πελάτη ένα προϊόν. Μετά έχουμε και κάποια άλλα πράγματα στο MIFID 2 για την προστασία των καταναλωτών. Σύντομα θα σας πω παραδείγματος χάρη υπάρχει μια διαδικασία διακυβέρνηση όπως λέγεται. Δηλαδή αυτός ο οποίος εκδίδει ένα προϊόν θα πρέπει να λέει ότι ταιριάζει σε ανθρώπους με αυτό το προφίλ, με αυτά τα κριτήρια, ήδη κατά τη διάρκεια της κατάρτισης αυτού του προϊόντος. Μετά θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στο κόστος ε, του προϊόντος. Και ένας άλλος ε, παράγων, ο οποίος ε, δεν αναφέρθηκε, είναι ότι έχουμε και τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και στην σχετική οδηγία του 2010 έχουμε προβλέψει ειδικά την ε, ΕΣΜΑ, την ε, Αρχή Χρηματαγορών και ότι αυτή θα ασχολείται με την προστασία των καταναλωτών. Η ΕΣΜΑ έχει ήδη λάβει πάρα πολλά μέτρα, παραδείγματος χάνει έχει εκδώσει οδηγίες για το πώς θα καταρτίζεται η δήλωση καταλληλότητας, δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της ε, πολλές ερωταποκρίσεις ε, για το πώς ακριβώς ε, μπορεί να ερμηνευθεί το κείμενο και το γράμμα του νόμου για να υπάρχει μια ομοιόμορφη εφαρμογή. Υπάρχει μια Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών στην ΕΣΜΑ, εκεί πέρα συναντώνται οι εθνικές αρχές εποπτείας αγοράς. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε κάνει αρκετά. Πρέπει επίσης να πω ότι ναι, πράγματι δεν μπορεί η Κομισιόν να εξετάζει την κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Η δουλειά μας είναι να εξετάζουμε αν η ευρωπαϊκή ε, νομοθεσία εφαρμόζεται σωστά στα κράτη-μέλη. Έχουμε λοιπόν δημιουργήσει πολλούς ε, μηχανισμού για τη βελτίωση της ε, προστασίας των καταναλωτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα λοιπόν έχει φτάσει η ώρα να ακούσουμε τους συναδέλφους. Κύρια μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να καλωσορίσω τους τρεις υποβάλλοντες στην αναφορά. Ε, η καταγγελία ξεκίνησε το 2012 με την αναφορά που είχατε υποβάλει τότε και μετά από ε, μεγάλη κινητοποίηση στους δρόμους της Γαλλικής και σε ολόκληρη την Ισπανία και της διεκδικής πολλών πλατφορμών γιατί αυτή η συλλογική απάτη, γιατί ήταν πραγματικά συλλογική απάτη, δεν ήταν μεμονωμένη περίπτωση, ήταν μια συλλογική απάτη που έπληξε ε, πολλές χιλιάδες Ισπανούς, κυρίως ηλικιωμένου ε, που νόμιζαν ότι έκαναν καταθέσεις των οικονομιών τους και δεν ενημερώθηκαν επαρκώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ε, ούτε βρέθηκαν λύσεις για να διορθωθεί η κατάσταση. Τότε η Ισπανική κυβέρνηση το 2012 ε, δέχτηκε τις απαιτήσει του Eurogroup ε, τον Ιούλιο του 2011 τότε αναφέρθηκαν ε, κάποια γραμμάτια προς τους μειωμένες εξασφάλισης κατόχους και τους κατόχους προνομιούχων μετοχών με ζημίες όμως της τάξης του 70% και το είπαμε στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη συνάντηση που είχαμε το 2003 με εκπροσώπους από όλες τις πλατφόρμες των θυγωμένων. Και τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή, αλλά ε, διαπιστώσαμε ότι έγινε μια προσπάθεια και ε, υποβλήθησαν νομοθετικές προτάσεις, αλλά παρόλα αυτά ε, η... δεν δόθηκε λύση για τους ανθρώπους που έχασαν τα χρήματά τους. Η Ισπανία τότε χρησιμοποιήθηκε ως πειραματόζω για την εκπόνηση σχετικής νομοθεσίας. Τελικά υιοθετήθηκε η Οδηγία 2014 59. Πρόσφατα, πολύ πρόσφατα όμως τέθηκε σε εφαρμογή η οδηγία αυτή. Και μάλιστα η, ε, σκληρότητα που δείχθηκε απέναντι στους ε, Ισπανούς ε, καταθέτες ήταν φρικτή. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ε, ήταν ιδιώτες που έκαναν καταθέσεις, δεν ήταν επενδυτές. Ενώ με τις τράπεζες ήμασταν πολύ συγκαταβατικοί, με τους πολίτες ήμασταν βάναυση μεγάλη αδικία που υπέστησαν αυτοί οι άνθρωποι. Επίσης, ε, μερικοί καταθέτες ήταν αγράμματοι, αναλφάβητοι και αναγκάστηκαν να υπογράψουν ε, α, καταχρηστικές πρακτικές, χωρίς καμία δήλωση καταλληλότητας χωρίς καμία συνδρομή άλλων προϋποθέσεων. Τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε ότι στην Ισπανία εφαρμόστηκε ένα νομικό καθεστώς που δεν είχε ακόμη τεθεί σε εφαρμογή. Αν το συγκρίνουμε με άλλες ε, χώρες, το, την 1η Ιουνίου του 2017 έγινε μια συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την τράπεζα Monte dei Paschi de Siena, ώστε με δημόσια κονδύλια επιτράπηκε στην ε, Ιταλική τράπεζα να ανακεφαλοποιήσει την τράπεζα με σεβασμό των ε, ευρωπαϊκών διατάξεων και ζήτησε από την τράπεζα αυτή να αποζημιώσει τους επενδυτές ε, ιδιώτες. Κάτι που δεν συνέβη στην Ισπανία. Γιατί στην Ιταλία έγινε η διάσωση με δημόσια κονδύλια, ενώ στην περίπτωση των τραπεζών της Γαλλικίας, με τη συνενοχή των κυβερνήσεων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που ακόμη είναι ε, κυβερνών κόμμα στη Γαλλικία, εξασ, ε, άφησαν στη μοίρα τους, στο έλεος των τραπεζών τους πολίτες. Δεν με ενδιαφέρει η ιδεολογία. Το θέμα είναι ότι οι κυβερνήσεις δεν στάθηκαν στο πλευρό των κατόχων των προνομιούχων αυτών, μετοχών που μόνο το όνομα έχουν προνομιούχες. Και δεν βοήθησαν τους πολίτες, τους άφησαν στη μοίρα τους, ανήμπορους τελείω και ανυπεράσπιστους. Τότε είχε σταλεί επιστολή στην Ισπανική κυβέρνηση. Θα πρέπει να σταλεί εκ νέου επιστολή στην κυβέρνηση της Γαλλικής και της, της Ισπανίας να μεριμνήσουμε για να δοθεί ένα αίσιο πέρα σε αυτή την κατάσταση και εμείς ε, ε, ζητήσαμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να καταθέσουμε νέα τεκμήρια, τουλάχιστον η δική μα πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στηρίζουμε φυσικά αμέριστα τις διεκδικήσεις αυτών των κατόχων των προνομίων μετοχών που κινητοποιήθηκαν ε, αλλά δυστυχώς χωρίς καμία δημόσια βοήθεια και στήριξη. Και όταν συζητήθηκε στη Γαλλικιακή Βουλή ε, αυτό το θέμα, ελάχιστη ήταν η υποστήριξη των τοπικών βουλευτών. Ε, η κυρία Ρόζα Φεραγκούτ, θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τους καλεσμένους μας, τους αναφερόμενους και να εξηγήσω ότι προσπάθησε να κάνει τότε η κυβέρνηση της Ισπανίας, η κεντρική, αλλά και η κυβέρνηση της Γαλλικίας. Γιατί μια και είμαστε στην προεκλογική περίοδο και θα έχουμε το Μάιο εκλογές, μερικές φορές ε, για ψηφοθερικούς λόγους επισκιάζεται την αλήθεια. Ας αφήσουμε λοιπόν τα κομματικά ιδεολογικά επιχειρήματα, σταθούμε σε πραγματικά περιστατικά και αδιάσυστα τεκμήρια. Όντως, στην Ισπανία, όπως και πολλές, σε πολλές άλλες χώρες, διατέθηκαν υβριδικά χρηματοπιστωτικά μέσα και μάλιστα προτάθηκαν μαζικά σε μικροκαταθέτες και μικροεπαιδητές που ήταν τα θύματα. Εξού και 22 αναφορές. Βέβαια από τους 22 αναφέροντες μόνο οι αναφερόμενοι από τη Γαλλικία εμφανίστηκαν εδώ, αλλά αναφορές υπήρχαν από όλε τις περιοχές της Ισπανίας. Μιλάμε για μέσα που διατέθηκαν μεταξύ το 2011, 2012 και 2013. Και μάλιστα είχαμε τη Συμφωνία της Βασιλείας το 2010 και την Ευρωπαϊκή Οδηγία το 2004, την πρώτη ΜΥΦΙΤ, που έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου και κατάλληλη επιτήρηση ώστε να μην ε, συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν έγινε τότε η σωστή επιτήρηση. Όταν ανέλαβε την κυβέρνηση ο Μαριάνο Ραχώη, το Λαϊκό Κόμμα, που ανέλαβε την κυβέρνηση της Ισπανίας το 2011-2012, αυτό που έκανε είναι να ανασκουμποθεί και να κάνει μια αναδιάρθρωση το 2012 όλων των τραπεζικών, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για να ε, εμποδίσει αυτή την ε, καταχρηστική πρακτική. Και μάλιστα ο κύριος Νουνιές Ήχο που ενοχλεί την κυρία Μιράντα πρότεινε ε, διαιτησίες στην Ισπανία, ώστε πάνω από, 75, πάνω από το 75% των υποθέσεων να διαθετηθούν με τη διαιτησία. Και μάλιστα συστήθηκε και μία, αποστο... μία επιτροπή παρακολούθησης που ενημέρωνε κάθε τρίμηνο το... την Βουλή. Και μάλιστα τροποποιήθηκε η νομοθεσία ώστε να μπορέσει το Ειδικό Ταμείο Εγγύης Καταθέσεων να βοηθήσει τους πελάτες, ώστε δύο στα τρία θύματα ανέκτησαν το 100% των ε, οικονομιών τους. Στη Γαλλική είχαμε 1.400, ε, 140.000 ε, καταγγελίες και 100.000 από αυτές διεκπαιρώθηκαν αισίως. Και μάλιστα είχαμε και συζήτηση στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου και το Κοινοβούλιο του 2015 κατέληξε σε ένα ψήφισμα που είναι ουσιαστικά το απάβγασμα όλων αυτών των συζητήσεων. Και όπως πολύ σωστά είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχαμε πρώτα την οδηγία του 2004, τη MIFID, μετά είχαμε τη δεύτερη οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων το 2008 και η μεταφορά αυτών των οδηγιών έγινε πολύ σωστά, όπως είπε ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ισπανία. Έχουμε τώρα το θέμα του, της τοπικής διοίκησης της Γαλλικίας. Στην αρχή ο Αλμπέρτο Νουνιεθιός ασχολήθηκε κυρίως με τους μικροκαταθέτες αυτούς. Προτάθηκαν κάποιες λύσεις και το, Ευρω... το Γαλλικιακό Ινστιτούτο Κατανάλωσης είχε εκατοντάδες χιλιάδες διαβουλεύσεις με πελάτες και μάλιστα οργανώθηκαν σεμινάρια ώστε όλοι να λάβουν τη σωστή ενημέρωση ε, είχαμε στενή συνεργασία με την εισαγγελία. Προτάθηκαν διαιτησίες και μάλιστα ήταν ε, ε, μια λύση που γενικεύθηκε στη συνέχεια στην Ισπανία και μάλιστα δύο στους τρεις καταθέτες ανέκτησαν στο έπακρο της οικονομίας τους στη Γαλλικία που ήταν υποδειγματική η κατάσταση και μάλιστα γινόταν 520 διαιτησίες την ημέρα την εποχή εκείνη και χρειάστηκε επάνδρωση των δικαστηρίων με επιπλέον προσωπικό στην Κορούνια και στο Βίγο, στη Γαλλικία, λόγω της έντασης του φόρτου των εργασιών λόγω των διατησιών. Και εκεί φάνηκε πόσο χρηστή ήταν η διακυβέρνηση στη Γαλλικία. Μπορεί να είχαμε κάποιες μεμονωμένες εξαιρέσεις, αλλά σε ό,τι αφορά τη διαχείριση που έγινε από την κυβέρνηση της Γαλλικίας και τη Βουλή της Γαλλικίας, αλλά και την κεντρική κυβέρνηση της Ισπανίας ήταν η υποδειγματική συνεργασία και η λύση των προβλημάτων ε, της συντριπτικής πλειοψηφίας των θεωμένων. Επίσης, ε, έχουμε δικαστές από το Βίγο και την Κορούνια που είπαν ότι ελάχιστες ε, υποθέσεις εκκρεμούσαν στα δικαστήρια. Πάνω από το 75% των υποθέσεων διευθετήθηκαν με διαιτησία και με ικανοποίηση των διαδίκων. Εγώ ζη, ζη, θα ζητούσα να, αρχιοθετηθεί, ε, να αρχιοθετηθούν οι αναφορές που είναι από το 2012, παρόλο που ξέρω ότι δεν υπάρχει συμφωνία, θα έπρεπε να το συζητήσουμε στους συντονιστές. Έγιναν πολλά, σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος και δεν θα ήθελα την περίπτωση αυτή να χρησιμοποιήσετε ψηφοθυρικά στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Εγώ είμαι στη διάθεση οποιοδήποτε θέλει βοήθεια αλλά θα ήθελα να διευκρινίσουμε ότι αυτά που ακούσαμε εδώ δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Καλή πρότασή σας ε, ότι είστε στη διάθεση ε, όποιων έχουν απορίες ε, και ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για προεκλογικούς λόγους αυτά τα σημεία, μόνο για ψηφοθυρικούς λόγους. Να δώσω τώρα το λόγο στους δύο υποβάλλοντες στην αναφορά για δύο λεπτά στον καθένα. Πρώτο ο κύριος Ροδρίγκης. Θα ήθελα να πω στην Επιτροπή ότι την πρώτη φορά που ήρθα εδώ, το 2013, Απρίλιο μήνα δεν κάνω λάθος, είχα φέρει έξι ντοσιέ γεμάτα έγγραφα και τα παρέδωσα στην Επιτροπή σας υπήρχε μια συλλογική αγωγή από 2.000 ε, πολίτες ε, και από το Γενικό Εισαγγελέα της Γαλλικίας. Ε, είχαμε συμβάσεις που δεν ήταν μόνο προσωπικές, αλλά καλύπτονταν από τη ΜΥΦΙΤ, παρόλο που δεν υπήρχαν ε, υπογραφές και μιλήσαμε για συμβάσει μετά το 2008. Η δική μου σύμβαση έγινε το 2010, όταν ήδη η τη λειτουργούσε εδώ και μερικά χρόνια. Επίσης, ε, ε, ήταν πολλές και διάφορες οι δικαστικές αποφάσεις. Έχουμε μια δικαστική απόφαση που κατηγορούσε την τράπεζα για καταχρηστική και δόλια πρακτική και για απάτη. Κατατέθηκαν αγωγές και έγιναν και μηνύσεις στην τοπική εισαγγελία και έγινε ανάλυση των καταγγελιών γιατί υπήρξαν καταγγελίες για απάτες. Επίσης, σας έστειλα αντίγραφα των ενημερωτικών δελτίων για τέτοιες επενδύσεις. Είχαμε μάλιστα ε, μερικά ενημερωτικά δελτία που ήταν 30 με 100 σελίδες. Πώς είναι δυνατόν ένας πελάτης ιδιώτης να διαβάσει όλη αυτή την τεκμηρίωση και να δηλώσει ότι τα κατάλαβε όλα με τους πίνακες, με τους ε, περίπλοκους μαθηματικούς τύπους και παρόλα αυτά λένε ότι ε, με τεκμηριωμένη γνώση έβαζαν την υπογραφή τους οι πελάτες. Ωραία όλα αυτά, ωραία η νομοθεσία, ωραία, ωραία στα χαρτιά, αλλά νομίζω ότι είμαστε πολύ καλόπιστοι. Η τράπεζα δεν κάνει πάντα καλά το έργο της και δεν αρκεί ε, η MIFID 1, αν το 2010 μου υποβάλλω μία πρόταση για, του, για τις προνομιούχες μετοχές με 1,5% επιτόκιο, όχι 7,4%. Μεταξύ του 2014 και το 2017 η κατάσταση δεν άλλαξε. Και σήμερα την ίδια κατάσταση την έχουμε με τις υποθήκες. Είναι μια δυναμική εσχροκέρδειας. Η Ισπανία δεν έχει τη κουλτούρα που έχουν οι σκανδιναβικές χώρες, παρόλο που μπορεί να πονάει αυτό που λέω μερικούς. Αν βρούμε ένα νόμισμα στο δρόμο, δεν την επιστρέφουμε σε αυτόν που το έχασε, αλλά το πατάμε για να μην το δει κανένας και το βάζουμε στην τσέπη μας. Τα καλά και συμφέροντα στην Ισπανία. Και το πρόβλημα δεν είναι με την ισπανική δικαιοσύνη, με μία-δύο δέκα αποφάσεις. Το είπε και η κυρία από το Λαϊκό κόμμα. Εκατό και χιλιάδες μας είπαν. Δεν είμαι μόνος μου. Το είπε η ίδια κυρία από το Λαϊκό Κόμμα. Εγώ δεν εκπροσωπώ εδώ κανένα πολιτικό κόμμα, ούτε με ενδιαφέρουν οι εκλογέ του Μαγίου. Εγώ ήρθα εδώ για να πω την αλήθεια. 500 ε, εκατομμύρια ήταν το χρέος της τράπεζας. Και το Εργατικό Κόμμα και το Λαϊκό Κόμμα χρωστούσαν χρήματα στην τράπεζα αυτή. Πλήρωσαν τα χρέη τους. Όλα αυτά τα όργανα, όλα αυτά τα κόμματα, όλες αυτές οι επιτροπές επέστρεψαν τα χρέη τους στην τράπεζα. Όχι. Και το 2009, όταν ο κύριος Φέχο υπέβαλε τα διαπιστευτήριά του στον Χουαν Κάρλος τον πρώτο, ρώτησε ο Χουαν Κάρλος, τι γίνεται με τις γαλλικιακές τράπεζες. Δεν έχω ιδέα λέει. Τότε αύριο να συναντηθεί με τον κύριο Φερνάντε Ορδόνιε, είπε ο Βασιλιά, που ήταν ο κυβερνήτη τη της ε, Ισπανική Κεντρική Τράπεζα. Τότε ο διοικητή τη Ισπανική Κεντρική Τράπεζα είπε ότι είναι σε τεχνική πτώχευση η Τράπεζα Γαλλικία. Και τι έκανε αυτό ο κύριο ένα χρόνο μετά. Δήλωσε ψευδός ότι η συγχώνευση αυτών των δύο τραπεζών θα είναι επικερδής. Και τότε είναι που καταβαραθρώθηκε ε, η αποταμίευση στη Γαλλικία. Αυτό δεν, είναι δεν είναι πολιτικό πρόβλημα, είναι πραγματικό πρόβλημα. Και τώρα την τράπεζα την, έχουν... την έχει αγοράσει μια τράπεζα της Βενεζουέλας. Δεν μας ενδιαφέρει η επιτήρηση, δεν αρκεί ο έλεγχος, δεν αρκεί η εποπτεία. Το διεθνέ Νομισματικό Ταμείο έχει κάθε 15 μέρες εκθέσεις από τράπεζες με προβληματικές πρακτικές. Πότε θα διορθώσετε αυτές τις αδυναμίες και τις ελλείψεις. Θα την πληρώσουν οι ιδιώτες καταθέτες. Αναλύστε την πολυσέλιδη τεκμηρίωση που σας έστειλα και μετά έλατε να μιλήσουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Ροντρίγκες, δύο λεπτά έχετε κι εσείς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι που αναφέρθηκε. Οι εκδόσει των μέσων, χρηματοπιστωτικών μέσων τη Κάισα Γκαλίσια και τη Κάισα Νόβα δεν έγιναν αργότερα. Μιλούμε για το 1988 από τους φορολογικούς παραδείσους, 2003, 2004, 2005, κυβερνήσεις Φράγκα και Ριβάρνε. Τις έχετε υπόψη. Και η μεγαλύτερη έκδοση έγινε το 2009 αμέσως μετά την ανάληψη ε, της κυβέρνησης της Γαλλικής από το ΕΛΚ. Οπότε δεν ήταν μεταγενέστερες αυτές οι εκδόσεις. Και αυτό για την ε, διάθεση των προνομίουχων μετοχών. Όταν λέμε ότι η διαιτησία είναι προσβολή, εννοούμε ότι οι τράπεζες αυτές που μας έκλεψαν, ε, ε, μέσω των μελετών καθοδηγούσαν και έλεγχαν τις διαιτησίες. Και για ένα ολόκληρο δεκάμινο οι διαιτησίες αυτές, οι διαιτητικές διαδικασίες δεν είχαν προκαθορισμένα κριτήρια. Οι διαιτησίες γινόταν αυθαίρετα. Μερικούς τους καλούσαν στην διαδικασία και άλλους όχι. Μερικές φορές ανάλογα με πολιτικές προτεραιότητες. Ουσιαστικά προτεραιότητες ε, εξυπηρετούσαν οι διαιτησίες. Ο κύριος Φίχο στις ε, συνεδριάσεις έλεγε «Αν κερδίσουμε τις εκλογές, τότε θα επιστρέψουμε τα χρήματα από τις προνομιούχες μετοχές». Ένα επιπλέον ψέμα, μία επιπλέον ψηφοθερική δήλωση. Επίσης, τα αποτελέσματα των διατησιών ήταν σαφή. Στην ε, Γαλλική επιστράφηκαν το 34% των χρημάτων με τις διαιτησίες. Αρχικά ήταν 5%, μετά έγινε 10%, έγιναν διαδηλώσεις, κινητοποίηση των πολιτών, συλλαλητήρια, έκλεισαν τα δημαρχεία, πολλαπλές κινητοποιήσεις και καταφέραμε χάρη σε αυτή την κινητοποίηση να φτάσουμε στο 30%. Μετά ε, έγινε το διάταγμα για την υποχρεωτική ε, επιστροφή που δεν προβλεπόταν στην αρχή και μετά είχαμε τις δικαστικές αποφάσεις μετά τις αρχικές στάσεις της Επιτροπής που μας έλεγαν ότι αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι <clears throat> να επιδιώξετε την ε, μεμονωμένη ακύρωση όλων των συμβάσεων, είτε δικαστικά είτε εξοδικαστικά. Και αυτό συνέβη στην Γαλλικία. Ε, με εξαίρεση 100 εκατομμύρια ανακτήσαμε το 90% των χρημάτων. Βέβαια, μία τράπεζα ε, διασώζεται με 9 δισεκατομμύρια, πωλήθηκε για 1 δισεκατομμύριο και ήδη από τον πρώτο χρόνο έχει κέρδη. Εξυπηρετώντα μόνο του μετόχου και όχι του πολίτε. Γι' αυτό μιλήσαμε για ασυμμετρία και άδικη μεταχείριση, γιατί οι μικροκαταθέτε μόνο εμπόδια βρίσκουν μπροστά του, ενώ οι ιδιωτικέ τράπεζε ε, ευνοούνται και λαμβάνουν ένα σωρό πλεονεκτήματα. Είδαμε τι συνέβη με τις προνομιούχε μετοχές. Εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσει για διαιτησία απορρίφθηκαν. Και στην έκθεση που μπορώ να σα υποβάλω, έχω πολύ περισσότερα στοιχεία. Ασύμετρη πληροφόρηση, αδικία ει βάρο των μικρών καταθετών, Δόλειε και καταχρηστικές πρακτικέ από τι τράπεζε που γίνονται για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που σας ανέφερα προηγουμένως. Και εκατομμύρια είναι οι θυγόμενοι ε, Ισπανοί Καλή η Μιφιντ 1, καλή και η Μιφιντ 2, αλλά τι γίνεται με τη μεταφορά της στο Ισπανικό Εθνικό Δίκαιο. Θα πρέπει να τραβήξουμε τα αυτιά των Ισπανικών αρχών. Δεν αρκούν οι οδηγίε και το είπε τη προάλλη η Υπουργό Οικονομία τη Ισπανία. Ότι το Ισπανικό οικονομικό θαύμα σήμερα βρίσκεται στα κάτεργα. Ευχαριστώ. Ε, Σα ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Νομίζω ότι είναι σαφές σε όλους ότι το, σύστημα είναι, το ζήτημα είναι αρκετά περίπλοκο και θα μας πάρει καιρό ακόμη. Πάντως, η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Αναφορών στο παρελθόν ήταν πολύ θετική και ε, νομίζω ότι βοηθήσαμε σε μεγάλο βαθμό να λυθεί ένα τμήμα του προβλήματος. Σταθήκαμε στο πλευρό των ε, υποβαλλόντων την αναφορά και οι δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν χρήσιμοι. Και ξέρω ότι οι υποβάλλονται στην αναφορά δεν έχουν μείνει ικανοποιημένοι από την κατάσταση και ζητούν ένα νέο γύρο συζητήσεων και αποζημιώσεων. Έχουμε πάνω από 20 αναφορές, μεμονωμένες αναφορές για το θέμα αυτό. Δύο μάλιστα δεν είναι καν ατομικές, είναι συλλογικές, έχουν, φέρουν πολλές υπογραφές. Αλλά θα πω κάτι για δύο ε, αναφορές δύο αναφεροντές αρνήθηκαν γραπτός ότι έχουν αποζημιωθεί είναι η 1761 του 2012 και η αναφορά 2228 του 2013 στην περίπτωση αυτή νομίζω λοιπόν ότι έχει κλείσει η περίπτωση και μπορούν να κλείσουν και οι δύο αυτές αναφορές. Στην περίπτωση των άλλων αναφορών είχα μόνο ένα αίτημα από την δική σας την πλευρά για να παραμείνει ε, ανοιχτή. Ε, δέχομαι την θέση αυτή και να αποστελούμε δύο επιστολές, ε, δύο επιστολές στην Ισπανία, στις αρχές της Γαλλικίας και του Βασιλείου της Ισπανίας να πω μόνο ότι παίρνω το θέμα στους συντονιστές για το αν θα κλείσει ή όχι. Βέβαια ότι είναι καλή ιδέα. Μάλιστα, λοιπόν, θα προστείλουμε δύο επιστολές στις ε, Ισπανικές αρχές και στις αρχές της ε, Γαλλικίας και ζητάμε όχι, όχι. Ε, δεν υπάρχει απαρτία. Το είπαμε και χτες. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε κάτι τέτοιο. το είπαμε χτες. Δεν έχουμε απαρτία. Ζητώ να πάρουν την απόφαση οι συντονιστές. Δεν έχουμε απαρτία. Μάλιστα. επί τη βάση του αιτήματός σας. Τι, θέλετε εσείς. Ε, θα ξαναδείξουμε το θέμα αυτό στο, Μάρτιο. Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα ένα μήνα πριν τις ισπανικές εκλογές. Ε, εγώ προτείνω να κλείσουμε αυτήν τη συζήτηση τώρα και να συνεχίσουμε μετά τις εκλογές, ε, αν το επιθυμείτε. Αν ε, θέλετε να ξαναγίνει ένας έντονος διάλογος ε, τον Μάρτιο στην Επιτροπή Αναφορών, έχετε δικαίωμα. Αλλά δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έλεγα εγώ είναι να είμαστε νόμιμοι, να τηρήσουμε τους κανόνες. Σύμφωνα με τους κανόνες υπάρχουν τρεις βουλευτές εδώ από μια επιτροπή 30 ατόμων. Η αριστερά λέει συνέχεια ότι πρέπει να έχουμε ε, απαρτία. Δεν μπορούμε να λάβουμε απόφαση. Η κυρία Μιράντα έφερε εδώ πέρα την αναφορά αυτή. Εγώ έχω μια πολιτική αξιολόγηση, η συνάδελφο έχει μια διαφορετική αξιολόγηση, πρέπει να πάει στου συντονιστέ. Να αποφασίσουν αν θα είναι ανοιχτή η επιτροπή, αν θα αποστείλουμε επιστολέ, αν θα ξαναπάει στην επιτροπή αλλά σύμφωνα με τους κανόνες. Δεν μπορούμε τώρα να λάβουμε απόφαση. Αυτό λέω. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Πράγματι δεν έχουμε απαρτία. Διακόπτεται τη διαδικασία λήψης απόφασης και θα ζητήσω από τη γραμματεία να το βάλει στην ημερήσια διάταξη των συντονιστών το Μάρτιο. Εντάξει. Παρακαλώ. Κοιτάξτε. Θα προσπαθήσω να τα πω ξεκάθαρα αλλά ευγενικά. Είναι πολιτική η συζήτηση. Έτσι. Το ε, ζήτημα αυτό μας απασχολεί από το 2012. Έτυχε να συμβεί τώρα. Ε, Εσεί τίποτα δεν κάνατε να το φέρετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε εσεί ούτε κανένα άλλο κόμμα. Εγώ μπήκα το Μάρτιο εδώ και από τότε που ανέλαβα καθήκοντα φρόντισα να μείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Εγώ κάνω τη δουλειά μου και εκτιμώ αυτό που είπε ο Πρόεδρο. Ότι το σημαντικό είναι να ακούσουμε του υποβάλλοντε την αναφορά. Γιατί δεν είναι ένα, είναι πολλοί και θα πρέπει να του ακούσουμε στέλνοντα επιστολέ γιατί δεν στοιχίζει τίποτα να στείλουμε επιστολή στην κυβέρνηση ζητώντα ενημέρωση. Αν μα επιβεβαιώσει η κυβέρνηση ότι όλα καλά, θα αρχιοθετήσουμε την αναφορά. Τι αναφορέ, μάλλον. Αν α, οι κυβερνήσει μα δώσουν ενδείξει ότι δεν υπάρχει επάρκεια αναφορά, θα πρέπει να συνεχίσουμε το έργο μα. Εγώ είμαι εδώ γιατί είμαι πολιτικό. Δεν είμαι παρατηρήτρια και δεν είναι κακό να είναι κανεί πολιτικό και ταυτόχρονα να υπερασπίζεται του συμπολίτε του κυρία Σταράς. Και θέλω να απαιτήσω λίγο σεβασμό, γιατί έχετε μία αιμονή, μία ιδεολειψία εις βάρος μου. Εγώ είμαι υπομονετική και θα είμαι και στο μέλλον υπομονετική, αλλά παρακαλώ ε, να το λάβετε υπόψη ότι χρήζουν σεβασμού οι υποβάλλοντες στην αναφορά. Θα ήθελα να μείνει ανοιχτή αναφορά. Είναι πολύ περιορισμένη, είναι δεμένα τα χέρια μου. Δεν μπορώ εγώ να αποφασίσω μόνος μου πρέπει να σεβαστώ τους ε, διαδικαστικούς κανόνες, τον εσωτερικό μας κανονισμό που προβλέπουν αυτά που είπε η Ρόζα. Να ζητήσουμε από τους συντονιστές να λάβουν την τελική απόφαση το Μάρτιο. Δεν έχουμε απαρτία τώρα. Και να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση αυτή για σήμερα. Δεν έχουμε τίποτα άλλο στην ημερήσια μας διάταξη. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία και σας εύχομαι καλό Σαββατοκυριακό. Εμείς θα συνεχίσουμε το Μάρτιο. Γεια σας.